Επειδή απουσιάζουν οι πρόεδροι και οι, και οι αντιπρόεδροι, οι υπόλοιποι, μου είπαν να το προεδρεύσω εγώ, αλλά αγγλιστή. Πρώτο θέμα έγκριση. Λοιπόν, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερον, Ανακοινώσει του Προέδρου. Η ΕΚΤ μας γνωστοποιεί ότι η συνεδρίασή μας της Δεπτέρας 8 Ιουλίου θα αρχίσει στις 2.30 το απόγευμα. Αυτό για να μπορέσει και ο κύριος Μάριος Ντράγκη να πάει αργότερα στη συνεδρίαση της Ευρωζώνης. Άλλη ανακοίνωση. On what? Market abuse. Α, για τις καταχρήσεις των αγορών. Έγινε λέει φοβερή πρόοδο στον τριμερή διάλογο και είναι φανερή ήδη η δυνατότητα συμφωνίας εάν το Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα ξεπεράσει ορισμένα προβλήματά του. Μήπως θέλει κανείς να δηλώσει τίποτε για αυτά. Όχι. Next uh, point. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο ετήσια έκθεση της ΕΚΤ του κυρίου Πιτέλα. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης είναι εδώ, ο κύριος Πιτέλα είναι. Έχει λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την Προεδρία σας. <laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Ευρωζώνη. Όπως ε, πολλοί από σας γνωρίζετε, το καθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε από το 0,6% η ε, ανεργία θα πλησιάζει απειλητικά το κατόφλι του 12%. Σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο οι αγορές αντέδρασαν πολύ νευρικά και η απόδοση των κρατικών ομολόγων των πιο ευάλωτων χωρών φτάσανε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ενώπιον αυτής της κατάστασης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενήργησε σωστά. Μάλλον, μάλιστα, επιτρέψατε μου να πω ότι πολύ καλύτερα από πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ω προς αυτό το τομέα λοιπόν θα πρέπει να χαιρετήσουμε ε, την θέση του, 2000, του Ιουνίου 2012 να μειωθούν ε, τα επιτόκια. Ε, τώρα, όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, το δεύτερο, η δεύτερη φάση επέτρεψε στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα να αναπνεύσει. Όμως όλα αυτά δεν άρκεσαν διότι οι ε, παραδοσιακοί μηχανισμοί μετάβασης της ε, νομισματικής πολιτικής ε, έχουν μπλοκαριστεί. Θέλουμε να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα κρατικών ομολόγων, το πρόγραμμα OMT. Η ανακοίνωση αυτού του προγράμματος σημάδεψε το σημείο καμπής για το 2012 γιατί επέτρεψε τη σταθεροποίηση των προσδοκιών των αγορών. Και ωστόσο η ενέργεια της έκτη δεν ήταν καθοριστική ούτε μπορούσε να είναι. Η κρίση, η κρίση μπορεί ανα πάσα στιγμή να αναζωογονηθεί, αναζωπηρωθεί όπως αποδεικνύουν οι διαφορετικές διαφορές ε, των spread. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά ζητήματα που αν δεν επιληθούν μπορεί να επιδεινώσουν την κρίση. Καθόμαστε στο χείλος ενός κρατήρα που κινδυνεύει να εκραγεί και το αίτιο αυτή τη κατάσταση είναι προφανέ προφανές κατά τη γνώμη μου. Η αδυναμία της εσωτερικής ε, ζήτησης που, καθιστά, που έχει καταστεί μάλλον πολύ αδύναμη λόγω των δογματικών πολιτικών λιτότητας και σταθεροποίησης. Για να διορθώσουμε όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην νομισματική πολιτική. Αυτές εδώ είναι οι δικές μου προτάσεις. Το πρόγραμμα OMT θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να έχει πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα, σήμερα ένα κράτος μέλος πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει τη στήριξη του Ταμείου Διάσωσης, ε, δηλαδή το κράτος αυτό θα υπόκειται σε πολύ αυστηρούς όρους ε, σε θέματα προπολογισμού. Ενώ αντίθετα θα πρέπει να αποσυνδεθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα OMT από αυστηρούς όρους σε θέματα πολιτικών δημοσιονομικών γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση. Είναι μια πρόταση ουσιώδης που θέλω εγώ να υποβάλω. Η κρίση που δυναμητίζει την Ευρωζώνη δεν είναι κρίση μόνο χρέους αλλά είναι ε, κρίση αδύναμης ζήτησης και αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη ζήτηση στις χώρες που έχουν δυσκολίες, δεν θα καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση. Οι πολιτικές λιτότητε που θα πρέπει να συνδεθούν με το πρόγραμμα OMT, με βάση αυτή την παράλογη αρχή των όρων της αιρεσιμότητας, θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την κρίση και αυτό φυσικά θα αντικατοπτρίζεται στο δημόσιο χρέος. Θα πρέπει λοιπόν, ε, κατά τη γνώμη μου, να αποσυνδεθεί η εφαρμογή του προγράμματος OMT από τις πολιτικές λιτότητας. Ε, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν στέκουν και δεν είναι τυχαίο που κανένα κράτος μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίησή του, γιατί ακριβώς κοινωνικά δεν μπορεί να σταθεί. Δεύτερο στοιχείο που θέλω να θίξω αφορά την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ε, και μέσω της ε, κεντρικής τράπεζας να στηρίζεται από την πραγματική οικονομία. Χρειάζεται περισσότερο θάρρος να διερευνηθούν νέοι δρόμοι, όπως η δυνατότητα να μειωθεί σε αρνητικά επίπεδα η deposit facility rate, για να αποφευθεί το ε, πιστοτικά ιδρύματα να ε, ασφαλίζουν τη ρευστότητά τους, δηλαδή να δανείζονται τα χρήματα από την έκτα και μετά να τα ξανακαταθέτουν στην ίδια τράπεζα. Και άρα τα χρήματα δεν, κατα... δεν κατέληξαν τελικά μέσα στην πραγματική οικονομία. Χρειάζεται δηλαδή από πλευρά τη ε, Κεντρική Τράπεζα μια μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία απέναντι στη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι διάφορε κοινότητε στην Ευρώπη καθώ ε, υπονομεύονται από την ανεργία και την κοινωνική, ε, τις κοινωνικές δυσκολίες. Θα πρέπει να σπάσουμε τα ταμπού, σεβόμενοι όμως τις συνθήκες. Θα πρέπει να σκεφτούμε τη δυνατότητα για την ΕΚΤ να αγοράσει asset-backed τη securities, έτσι ώστε να δώσει μεγαλύτερη ρευστότητα στην οικονομία. Για αυτό το θέμα νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε η αγορά τέτοιων asset-backed securities να οδηγήσει στο να τροφοδοτήσει νέες φούσκες. Επίσης δεν θα πρέπει η έκτη να γεμίσει αμφίβολης προέλευσης ε, ε, ομόλογα απειλείται η σταθερότητα Ολόκληρη τη Ευρωζώνης και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε με περισσότερο θάρρος στην Τραπεζική Ένωση. Χάρη στην καθοριστική συμβολή της Επιτροπής μας και του Ευρωκοινοβουλίου, το 2012 τέθηκαν οι βάσει για να υλοποιηθεί το ενιαίο σύστημα τραπεζικής εποπτείας όπου επικεφαλής θα είναι η ΕΚΤ. Η απόδοση, ανάθεση μάλλον τη εποπτείας όλων των τραπεζών στην ΕΚΤ ε, δίνει στην ε, κεντρική μας τράπεζα μια ε, τρομερή δύναμη, τρομερή εξουσία που θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από μεγαλύτερη ευθύνη και διαφάνεια. Ο κανονισμός για το ενιαίο σύστημα υποπτίας που είναι υπό έγκριση περιλαμβάνει σημαντικέ δημοκρατικέ ρήτες όπω η έγκριση από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου, του διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εποπτείας, κανόνε οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσει συμφερόντων. Η ε, νομοθεσία αυτή που είναι υποδιαπραγμάτευση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις και κυρίως αναφέρομαι στην ανάγκη να επιτευχθεί η δημοσίευση των πρακτικών του Συμβουλίου Εποπτείας. Το 2012 μας έφερε σε μια έκτα πολύ πιο ισχυρή που μπορεί όμως να ενσταθεί πιο θαραλέα στο πεδίο των μη συμβατικών πολιτικών. Αυτή η θεσμική ισχύ θα πρέπει τώρα να συνοδευτεί από μεγαλύτερη ευθύνη και διαφάνεια. Γιατί οι πολίτες ε, και εμείς που τους αντιπροσωπεύουμε έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε πώς διαχειρίζεται η τράπεζα αυτές τις πολιτικές και αυτά τα σημαντικά μέτρα ακριβώς προς χάρη του παρόντος και του μέλλοντος της κοινότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Θα ήθελα να θυμίσω όμως ότι πρόκειται για την ετήσια έκθεση για το 2012, έτσι, επί αυτού του έτους είναι η ετήσια έκθεση. Δεν αφορά ακόμα την Τραπεζική Ένωση. Έχουμε άλλες εκθέσεις που μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο στο σκιώδη συγγητή, στη σκιώδη η συγγήτρια από το ΕΛΚ είναι η κυρία Γκολτ Πέλτς. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όσα έχει κάνει και να μιλήσω για το γενικότερο πλαίσιο. Πρώτον, αφού μιλάμε για την ΕΚΤ, από τη δική της πλευρά πρέπει να δούμε τα πράγματα. Άρα, πιστεύουμε ότι θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα καθήκοντα της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ έχει συγκεκριμένο ρόλο στον οικονομικό τομέα, στην οικονομική σφαίρα και φυσικά αυτά αφορούν και την απασχόληση, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δεδομένων αυτών που αφορούν την απασχόληση και την ανεργία και της δουλειάς της ΕΚΤ καθεαυτήν. Λοιπόν, για τη γνωμοδότησή μου τώρα. Τη δομή της έκθεσης την εγκρίνω. Νομίζω ότι είναι καλό που θίγει όσα θίγει για την Τραπεζική Ένωση και την νομισματική πολιτική. Για αυτή την τελευταία το πιο σημαντικό για μένα θα ήταν ότι επειδή συμφωνούμε ότι η μείωση των επιτοκίων είναι καλό πράγμα, να το αναφέρουμε ως θετικό στοιχείο της έκθεσης, να το τονίσουμε περισσότερο, καθώς και άλλα, άλλες πτυχές της νομισματικής πολιτικής. Δεν είμαι τελείως βέβαιη, αλλά ίσως να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα και με τους υπόλοιπους σκιώδεις, το πώς δηλαδή, το πώς δηλαδή θα μπορούσαν να αυξηθούν τα κονδύλια που αφιερώνει η έκτες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δεν συμφωνώ όμως με την προσέγγιση που θα ήθελε Amit érdekesnek és jónak is tartok, hogy kimondja a jelentés. Την αλλαγή που προβλέπει εδώ για το OMS. Τα νομισματικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ έχουν εξαντληθεί πια και γι' αυτό θα έπρεπε να προσπαθήσει να βρει και άλλους δρόμους και άλλα εργαλεία και μεθόδους μέσα βέβαια στα πλαίσια της εντολής της. Δεν νομίζω ότι η αναθεώρηση του καταστατικού της όμως είναι απαραίτητη ως προς τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της πλήρους απασχόλησης. Η πλήρης απασχόληση για μένα είναι κάτι αμφισβητήσιμο η προσέγγιση που βασίζεται δηλαδή στην πλήρη απασχόληση. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνεται δημοκρατικά ο νομισματικός έλεγχος και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της τράπεζας, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει αυτό δικαιολογία για την έλλειψη διαφάνειας. Τώρα για τα συναλλάγματα πιστεύω ότι αυτά έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, την ισοτιμία του ευρώ δηλαδή. Και ένα λανθασμένο επιτόκιο θα είχε πολύ αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη. Για την Τραπεζική Ένωση συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση αν και το θέμα αυτό το θεωρώ λεπτό. Πρέπει να συμβαδίζει η συζήτησή του, να συνοδεύει τη δική μας συζήτηση των γενικότερων πτυχών της Τραπεζικής Ένωσης. Για μένα υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ. Όχι μόνο αυτής της ετήσιας έκθεσης αλλά σε όλες. Είναι δεύτερη φορά δυστυχώς που μπορώ και πρέπει να επαναλάβω το ίδιο. Ότι η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν δίνει καμία σημασία στα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι βουλευτές. Αγνοεί απολύτως τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Αντίθετα δηλαδή από αλληλοβοήθεια οι μεν δυσκολεύουν τη δουλειά των δε. Γίνονται εκθέσεις, γράφονται συστάσεις και τις αγνοούν απλώς στην ετήσια τους έκθεση. Άρα συμφωνώ με τη δομή και το γενικότερο περιεχόμενο, αλλά έχω αυτή την αντίρρηση και θα καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίλ Τόρβαλτς, αλλά έχω την εντύπωση ότι απουσιάζει. Από τους φιλελευθέρους ποιος θα αντικαθιστά, υπάρχει κανείς. Ουδής. Καλώς, πράσινη. Ο κύριος Μπεσέ έχει το λόγο από τους πρασίνους. Ah, Κύριε Φιλίπ Ραμπρέξ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Α, εσείς είστε στη θέση του κυρίου Μπασέ. Για να είμαι ειλικρινή, είστε κυρία Εύα Ζολή. Ξέρω ότι δεν είμαι στο ύψο της, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό είναι το gender mainstreaming από την ανάποδη όμως. Να μιλήσει και κανένα άντρα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, Ευχαριστώ τον κύριο Πιτέλα για την αρχική του έκθεση. Θέλω να επικεντρωθώ σε μερικά σημεία μόνο, ε, στα οποία θα επιθυμούσαμε εμείς να προσθέσουμε μερικά πράγματα. Περί τίνος πρόκειται. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι βεβαίως κεντρική τράπεζα, αλίμονο. Αλλά ε, δεν θα πρέπει να γνωρούμε ότι την επιφορτίζουμε και με άλλα θέματα όπως είναι η Τραπεζική Ένωση και η Εποπτεία. Επίσης δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι αυτό τον καιρό γίνονται συζητήσεις και μάλιστα πολύ ε, σκληρές πολλές φορές μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων έτσι ώστε να υπάρχει ένας γερός όσο και παρκής ε, δημοκρατικός έλεγχος στην τράπεζα στα πλαίσια αυτών των ευθυνών της. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ε, σωστό να το παραγνωρίσουμε αυτό στην ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα είχε κάτι νοσηρό αν δεν το κάναμε Αφήστε δε που θα επαρεξηγεί το κιόλας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ, ε, είναι τμήμα αυτού που συχνά αναφέρουμε αυτό το πραγματάκι που το λένε Τρόικα και έχει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα στις χώρες που είναι σε προγράμματα, δηλαδή μνημόνια. Ο ρόλος της ΕΚΤ και εδώ μέσα είναι λίγο περίεργος διότι υπερβαίνει κατά πολύ την νομισματική πολιτική και θυμίζω ότι η ε, συνθήκη μπορεί να δίνει πλήρη ανεξαρτησία και αδιαπραγμάτευτη στην ΕΚΤ για την νομισματική πολιτική αλλά δεν ισχύει και το ίδιο για τα υπόλοιπα καθήκοντά της. Όταν λοιπόν λειτουργεί ως μέλος της Τρόικα η ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα ή συνεισφέρει στη λήψη τους που δεν έχουν μεγάλη σχέση με την νομισματική πολιτική. Γι' αυτό θα πρέπει ρητά να αναφέρεται πιστεύω πιστεύουμε εμείς σε αυτό το ρόλο. Και θυμίζω την ε, πρόσφατη ε, διένεξη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι γνωρίζουμε ότι, αν δεν είχε ότι δεν κουρεύτηκε από την αρχή το ελληνικό χρέος από το 2010 είναι επειδή τα είχε στυλώσει, για να το πω έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, και θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθεί αυτό. Επίσης, ε, συμφωνούμε ε, για τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές σε μεγάλο βαθμό με αυτά που λέγει ο εισηγητής. Υπάρχουν μερικά στοιχεία ενδεχομένως που θα μπορούσαμε να δούμε στην προοπτική αυτή πώ έχει η κατάσταση των κρατών μελών που επιθυμούν να βγουν από τα προγράμματα βοήθειας, οικονομικά προγράμματα ή μνημόνια. Επίση, να πω δύο λόγια για την Ιρλανδική ιστορία των Promissory Notes ε, για το πρόγραμμα ΕΛΑ της επίγουσας βοήθειας δευστότητας θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, ε, ότι έχει κάνει πρόοδους η ΕΚΤ για το μηχανισμό επίγουσας ενίσχυσης μορφή ρεστότητα. Θα πρέπει όμως να το προχωρήσουμε και να αναγκάσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας ανακοινώσει ποια ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει βοηθήσει ένα χώρα και με ποια επιτόκια σε αυτή την πίστοση που τους έχει ανοίξει. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη διευκρίνηση στα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το asset back securities, δηλαδή ε, οι εγγυήσει που κατατίθενται από τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή αν μη τι άλλο ανακατηγορία στοιχείων ενεργητικού για να ξέρουμε με ποιο τρόπο έρχεται να τα αξιολογήσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, θέλαμε να ε, προσθέσουμε μια ρητή αναφορά για τις μυστικές συμφωνίες για ε, net financial assets μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών και της ΕΚΤ που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα ποσά ανακατηγορία στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή και, και ομόλογα συγγνώμη κρατικά, ε, που διαθέτει κάθε κεντρική τράπεζα και που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ε, διακρατούν. Και επίσης θα θέλαμε να φέρουμε και κάποια στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί ή όχι να εθαρρύνει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν δεν έχει χρόνο ενδεχομένως η Εύα να ασχοληθεί με αυτά η Εύα να λαμβάνω ευχαρίστω στην έκθεσή της Σκιώδης. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Έπινγκ των συντηρητικών που είναι Σκιώδης ηγητής επίσης για την ομάδα του. Um, thank you, Madam President. First of all, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πιτέλα για το σχέδιο εκθεσής του, το οποίο πηγαίνει πολύ πιο πέρα βέβαια από αυτά που δέχεται η ομάδα μου, ωστόσο είναι πολύ σαφής, ακόμα και να ακολουθεί τη λάθος κατεύθυνση. Ο εισηγητής επενεί τα LTRO, ε, δεν είναι, είναι μάλλον κατά των ε, δεσμεύσεων ή των όρων για τα όμικρον νη σίγμα κτλ. είτε για, κατά των ενέσεων ρευστότητα, κατά της χρήσης του συστήματος επίγουσας ε, ενίσχυσης υπομορφή ρευστότητα, Όλα αυτά δείχνουν προς μία κατεύθυνση κύριε εισηγητέ, τα, ότι δηλαδή το να βγάλουμε φρέσκο χρήμα είναι η μόνη λύση για, τις, ε, τις, για να ρίξουμε τις τιμές για να σώσουμε την οικονομία. Τέτοιο φρέσκο χρήμα δεν καλύπτεται από την δημιουργία οικονομικής αξίας. Το αποθεματικό είναι η ε, εξάρτηση από φθηνό χρήμα και όχι οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία όπως θα έπρεπε. Και κατά σύμπτωση αυτό το Σαββατοκυριακό η Τράπεζα Διεθνών ε, ε, Διατησιών επέκρινε αυτή την προσέγγιση που επιτρέπει την αναβολή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και να παραθέσω, κυρία Πρόεδρε, τη διατύπωση αυτής της έκθεσης ε, διεθνών, ε, διεθνούς διατησίας που λέει ότι γίνεται όλο ένα και πιο ξεκάθαρο πως οι κεντρικές ε, τράπεζες δεν μπορούν να κάνουν ό,τι πρέπει για να ενισχύσουν τις αδύναμες οικονομίες και να επιστρέψουν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι στιγμή η συνέχιση των χαμηλών επιτοκιών και των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών έχουν καταστήσει πιο εύκολο για το ιδιωτικό τομέα να αναβάλει την μόχλευση και ευκολότερο για τις κυβερνήσεις να αναβάλουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Εν γέννη, Πρόεδρε, πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε μάλλον επικριτικοί και να έρθουμε σε περισσότερη λογική ρεαλιστική σε αυτή τη συζήτηση και την έκθεση και προς αυτό το στόχο θα υποβάλω διάφορες τροπολογίες και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να δουλέψουμε επικοδομητικά για την εξέφραση συμβιβασμών. Ευχαριστώ. Δύσκολο θα είναι όμως δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν. Τώρα δεν έχω άλλους σκιώδεις γιατί η Γκούδε δεν μας δήλωσε κανέναν. Περνάμε στους υπόλοιπους που ζήτησαν το λόγο. Πρώτα ο κύριος Χουάν Γκιόγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτον μια αντίδραση σε αυτά που είπε ο κύριος Έπινγκ. Τις ίδιες επικρίσεις θα τις έκανε και για την τράπεζα της Αγγλίας που κάνει quantitative όσο θέλει. και που κάνει ακριβώς αυτά που κατηγορείται, αλλά που καταφέρνει να διατηρήσει ένα κλίμα όπου υπάρχουν χαμηλά επιτόκια, όπως και η ΕΚΤ, που είπε και ο κύριος Πιτέλα, διατηρεί ακριβώς τα επιτόκια σχετικά χαμηλά. Έρχομαι στην έκθεση του κυρίου Πιτέλα τώρα. Αντίθετα από άλλους βρίσκω ότι τονίζει ακριβώς τα θέματα που πρέπει να θίξουμε και εμείς οι βουλευτές στην τράπεζα, προς την τράπεζα και που αρχίσαμε ήδη να τα θέτουμε στον νομισματικό διάλογο. Έχει δίκιο που τονίζει ιδιαίτερα την έλλειψη δημοκρατίας στα νομισματικά. Δύο παραδείγματα. Το πρώτο, ακριβώς αυτή η εξαγορά των δημοσίων χρεών. Όλοι τονίσαμε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει πολύ μεγάλα τμήματα του ελληνικού και του πορτογαλικού χρέους και σε κάθε διάλογο ερωτούμε τον κύριο Ντράγκη. Κερδίζει η ΕΚΤ από τα χρέη αυτά. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεύτερον, που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πράγματι όταν η ΕΚΤ βάζει χρήματα στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα και μάλιστα με περισσότερους τίτλους από ό,τι πριν, τότε τίνει να γίνει ένα αρνητικό στοιχείο που επιτρέπει τελικά στις ιδιωτικές τράπεζες να συνεχίσουν την κερδοσκοπία. Και θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής της τράπεζας. Τέλος, οι ισοτιμίες που δεν την χάνουν καμία απολύτως συζήτηση ενωσιακώς. Και άρα αυτό που γίνεται τελικά είναι ότι συμφέροντα μισοκριμένα ορισμένων χωρών που υποστηρίζονται από την, που ωφελούνται από την τωρινή πολιτική γιατί ξέρουμε ότι η πολιτική του σκληρού ευρώ προς το δολάριο ωφελεί χώρες που έχουν αποθέματα, πλεονάσματα όχι λόγω της ανταγωνιστικότητάς τους ως προς τις τιμές, αλλά της ανταγωνιστικότητας εκτός τιμών, πέρα από τις τιμές. Άλλες χώρες αντίθετα χρειάζονται ένα πιο αδύνατο νόμισμα που να τους επιτρέψει να αντισταθούν στον ανταγωνισμό από τις χώρες της δολαροζώνης. Και αυτό δεν το συζητάει η ΕΚΤ, όχι μόνο γιατί δεν είναι δικό της θέμα επισήμως, αλλά δεν συζητιέται ούτε και από το Συμβούλιο Υπουργών, Υπουργών Οικονομικών, το οποίο μπορεί να ζητήσει από την ΕΚΤ, που έχει τα κατάλληλα εργαλεία, να εφαρμόσει άλλη πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε και ο κύριος Πιτέλα έχει δίκιο που τα θέτει. Ευχαριστούμε πολύ. Αν είχα το λόγο θα σας ρωτούσα το εξή. Θα σας δίνω να το εξή. Το να είναι κανείς ανεξάρτητος δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και αντιδημοκρατικό. Βέρνερ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διάβασα την έκθεση και άκουσα τα σχόλια του κυρίου Πιτέλα. Πολλά από αυτά που λέει είναι σωστά, αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία που δεν μπορούμε να τα δεχτούμε χωρίς συζήτηση τουλάχιστον. Ορισμένα αμφιλεγόμενα θέματα δηλαδή. Πολύ συνοπτικά στο σημείο 10 θεωρεί ε, α, να κοιτάξουμε τις συνθήκες και το καταστητικό για ε, να ε, είναι δύο ισότιμοι στόχοι η σταθερότητα του νομίσματος και των τιμών. Ε, ναι, αυτή είναι μια ιστορία που δεν έχει να κάνει ε, παρόδο με το καταστατικό, είναι επί της ουσίας. Ποια είναι η σωστή νομισματική πολιτική για το μέλλον. Γιατί εδώ και δεκαετίες γίνονται συζητήσεις, ακόμα πριν έρθει το ευρώ, και αυτό απαιτεί ε, ουσιαστική αλλαγή των συνθηκών, αναθεώρηση και τροποποίηση, όχι κάποιες μικροαλλαγές και προτάσεις. Το πολύ πολύ να είναι συντακτική συνέλευση αν δεν είναι αναθεώρηση. Δηλαδή το σημείο 10 δεν μπορώ να φανταστώ ότι το διεκπεραιώνουμε έτσι εμπαρόδο, διότι ε, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και καλά θα έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλά κάνει να τηρεί τον νόμο και το δίκαιο. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε την παράγραφο 12. Καλή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κοιτάξει περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις ε, της πολιτικής λιτότητας στα κοινωνικά, στο Α και στο Β. Τι δουλειά έχει εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν κάνει οικονομίες και περικοπές η τράπεζα, οι κυβερνήσεις το κάνουν. Δεν φταίει η Κεντρική Τράπεζα που έχουν υπερχρεωθεί και έχει πάει το χρέος των κρατών σε τέτοια δυσθεώρητα ύψη. Το πολύ πολύ μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αν δω την ετήσια έκθεση ε, για την Τράπεζα της Βασιλείας των Διεθνών ε, Διακανονισμών που είναι η οργάνωση των 19 ηγετικών κεντρικών ε, τραπεζών παγκοσμίως και κρατών. Εκεί τη ζητείτε. Η τράπεζα αυτή στην ετήσια έκθεση θα πρέπει να διαπιστώνει ότι το φτηνό χρήμα σε οθεί προς τη χρέωση αντί προς τις οικονομίες και αναχώρα διαφέρουν οι καταστάσεις και οι πρόοδοι που γίνονται. Και αλλού γράφει στο δεύτερο τμήμα, στην έκθεση Πιτέλα, για τα χαμηλά επιτόκια. Τα χαμηλά λοιπόν επιτόκια οδηγούν σε επιθετική ανάληψη ρίσκου και δημιουργούν ανισορροπίες όσο και στρεβλώσεις των τιμών στις χρηματαγορές. Και πιστεύω ότι βάσει της παρούς ετήσιας έκθεσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική, η, μάλλον η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έχει αλλάξει τακτική. Αυτό δεν ε, Αρέσει στους κερδοσκόπους, αλλά τις πταίει. 9,5 9,5-3 είναι το χρέος στην Ευρώπη, 2,8 το ε, ΑΕΠ. Ε, κάποια στιγμή φτάνουν και στα όρια μας. Δεν μπορεί να καθίσταται υπεύθυνη για τα πάντα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το είπε ήδη ο πρόεδρος, η Τραπεζική Ένωση είναι εν το γεννάστε ακόμα δεν έχει γίνει ούτε είναι αντικείμενο της ετήσιας έκθεσης του 2012 γιατί εκεί οι πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Ε, αλλά αν θέλετε να το κάνετε σε αυτό, ε, σε μια έκθεση μπορεί να γίνει στραμμένη προς το μέλλον, θα πρέπει να μπει στη σωστή του διάσταση. Κύριε Πιτέλα, είπατε και γράψατε ότι είναι ένας θαραλέος δρόμος προς την Τραπεζική Ένωση να επιφορτιστεί κεντρική τράπεζα με την εποπτεία όλων των τραπεζών. Μα γεγονό είναι ότι είναι μεγάλες τράπεζες με ένα ισολογισμό πάνω από 30 δισεκατομμύρια και υπάρχουν και μεγάλες νομικές επιφυλάξεις είναι οι δύο μεγαλύτερε τράπεζε ε, σε κάθε χώρα. Λοιπόν, είναι τεράστιε οι επιφυλάξει για την ανάληψη του συνόλου των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη Εποπτεία. Και στη Γερμανία τουλάχιστον τον τελευταίο λόγο έχει το Συνταγματικό Δικαστήριο. Και έγινε εκεί μια ακροματική διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε, σε αντίθεση με το πρόγραμμά τη μέχρι τώρα, ότι ε, αυτό το απεριόριστο ε, στην ε, παροχή που έχει θα το περιορίσει γιατί υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Και ε, σε ό,τι αφορά το κρατικό χρέος, ο διαχωρισμός των τραπεζών από τα κράτη δεν ξεπεράστηκε από το πολύ φθηνό χρήμα. 1% ήταν τα επιτόκια τα διατραπεζικά ε, και οι τράπεζες αυτές αγόραζαν κρατικά ομόλογα με επιτόκιο 6% και αυξήθηκε κατά πολύ η εξάρτηση και η τράπεζα για τους διεθνείς διακανονισμούς ε, λέγει ότι τα κρατικά ομόλογα έχουν μηδενικό ρίσκο. Εξακολουθεί να το πρεσβεύει αυτό. Θα πρέπει να έχουμε εδώ το θάρρος στην Επιτροπή μας να λέμε τα κρίσιμα πράγματα πέρα από το νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρό τους και να μην έχουμε ένα ευχολόγιο τώρα ε, για, ως γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση που είναι για το 2012. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλους αγεγραμμένους ομιλητές. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Ο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους ε, που πήραν τον λόγο για τις παρατηρήσεις τους, ε, για τη στήριξη αλλά και για τις ε, επικρίσεις και για τις πιο επίμαχες ερωτήσεις που έθεσαν. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Υπάρχουν θέματα για τις οποίες θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει να φτάσουν χρήματα, τα χρήματα της ΕΚΤ κατευθείαν στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να εμβαθύνουμε φυσικά. Εγώ εδώ έβαλα ένα κεφάλαιο που πέρυσι δεν υπήρχε για τις πολιτικές συναλλαγές, συναλλαγματικών ισοτιμιών. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα και είναι σίγουρο ότι θα είναι αντικείμενο προβληματισμού. Εγώ είμαι απόλυτα διαθέσιμος για τους κοιόδης και για όλους τους συναδέλφους για να ορίσουμε μαζί ε, σημεία ε, κοινά συνένεση. Η ΕΚΤ ε, έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο ένας εξαιρετικά ισχυρός θεσμικό φορέας και είναι σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο να βρει σε αυτή την υπόθεση μια θέση κοινή, συνενετική. Από πλευρά μου λοιπόν έχω απόλυτα τη διάθεση να λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις που θα γίνουν και θα υπογραμμιστούν και από τους συναδέλφους και σε αυτή τη φάση που προηγείται της παρουσίασης των ε, τροπολογιών, αν οι συνάδελφοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μου, είμαι απόλυτα διαθέσιμος. Ευχαριστώ σας και εγώ σας ευχαριστώ. Και το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η προθεσμία που έχει προταθεί για τις τροπολογίες είναι η 10η Ιουλίου. Οι τροπολογίες αυτές θα συζητηθούν εδώ στις 23 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει 4 ή 5 Νοεμβρίου και ολομέλεια ενδεικτικός προγραμματισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή για το Δεκέμβριο. Δέχεστε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία λοιπόν για την υποβολή των ε, τροπολογιών η 10η Ιουλίου. Περνώ στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Μπούρκαρντ για την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετωνία, την προσχώρηση της Λετωνίας στο ευρώ, το έχουμε ήδη συζητήσει και σήμερα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και μετά θα ψηφίσουμε. Κύριε Σιγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριο Μπάλτς, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, πολύ για τις τροπολογίες που κάνατε. Γενικώ συνολικά ήταν 22 αυτές που κρατήσαμε και ε, συμφωνήσαμε και πρέπει να σας πω ότι ήταν και πολύ μικρή προθεσμία, 24 ώρες. Αλλά παρόλα αυτά οι συνάδελφοι βρέθηκαν για να κάνουν τροπολογίες. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να πω και λόγω και της γνωστής αφορμής ήταν πολύ ε, περιορισμένη η χρονική δυνατότητα ε, που είχαμε και το περιθώριο λόγω του κατεπήγοντος και σήμερα ήταν η μόνη ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε τροπολογίες και να ψηφίσουμε αμέσω μετά για λόγους χρονικούς. Αυτό το γνωρίζετε, το έχουμε γράψει και αυτό στην έκθεση ότι ήταν πάρα πολύ σφιχτά τα χρονικά περιθώρια. Πρέπει να πω ότι γενικά χάρηκα πάρα πολύ που δεν χάθηκε καμία τροπολογία και εγκρίθηκαν όλες. Ναι, Βέρνερ, υπάρχουν και τέτοια πράγματα, λέω στον κύριο Λάγκεν. Και γενικά ήταν ε, θετική η ε, αντιμετώπιση απέναντι στην είσοδο της ε, Λετωνίας στο ευρώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους και για τον επικοδομητικό διάλογο της περασμένης εβδομάδας και συμφωνήσαμε με τους κοιόδης ηγητές σε ορισμένες τροπολογίες να τις ομαδοποιήσουμε και να τις συνοψίσουμε, διότι κατά την άποψή μας έβαιναν προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες, και Τελικά ε, πιστεύω ότι φτάσαμε σε ένα καλό θετικό αποτέλεσμα και 7 συμβιβαστικές συνολικά. Επίσης, στις τροπολογίες εδώ κάναμε κάποιες προτάσεις και τις εγκρίναμε στο συμβιβασμό α, β, ε και f. συμβιβασμοί C και G ε, διευρύνουν κάπως το πλαίσιο της έκθεσης σε μερικά στοιχεία και όπως είδαμε και ζητήθηκε και την περασμένη εβδομάδα και έγιναν και τροπολογίες που ε, αφορούν την εξάρτηση ε, από ενέργεια και το θέμα των τιμών ε, βάλει σε ένα συμβιβασμό υπαριθμών D. Ε, Επίσης ε, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που αποφασίσαμε συνειδητά να μην τα βάλουμε στην έκθεση. Το μόνο θέμα που μας απασχολεί είναι η ένταξη της Λετωνίας στην Ευρωζώνη και δεν έχει απαραίτητα νόημα να επεκταθούμε σε άλλα θέματα. Στην τελευταία συνεδρίαση, την Πέμπτη των σχεδόν συντονιστών, αποφασίσαμε να ζητήσουμε κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ξανασκεφτεί ε, τα κριτήρια σύγκληση, να μην αποφασίσαμε αυτό απ' έξω. Θεωρούμε και πάλι σκιώδη ότι δεν είναι εντό θέματο, γιατί και στην τελευταία προσχώρηση, πριν από μία διετία η Αστονία, θα θυμάστε, ε, ακούστηκε αυτή η επίκριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει. Το υποστηρίζω και εγώ και το είχα πει και στη συζήτηση που έγινε των σκιωδών. Τα κριτήρια σύγκλησης θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε, να τα ξανασκεφτούμε για να μην πω να τα αναθεωρήσουμε. Ε, να βρεθεί όμως το αντίστοιχο, το σωστό πλαίσιο, όχι σε αυτή την έκθεση. Θα το καλωσόριζα επίσης εάν συμφωνούσατε με αυτή μου την τοποθέτηση. Και τέλος θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να πω ότι καταβάλαμε προσπάθεια να διατηρήσουμε τη θετική στάση της έκθεσης και την ευνοϊκή και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά. Ε, με ενίσχυσαν και οι τροπολογίες την άποψή μου ότι η Λετωνία θα είναι ένα νέο ευπρόσδεκτο μέλος στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει Πρόεδρος, και δίνω το λόγο στους Σκιώδης. Σοσιαλιστές, ο κύριος Κούτας. Thank you, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι και εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα με τον κατάλογο ψηφοφορίας και εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά ότι θα υπερψηφίσουμε την ένταξη της Λετωνίας στην ε, Ευρωζώνη. Χαίρομαι που ο εισηγητής βρήκε και μια λύση για τα πολιτικά προβλήματα που υπήρχαν ακόμη. Μεταξύ άλλων και στις τροπολογίες αναφέρομαι για την αναθεώρηση των κριτηρίων σύγκλησης και την εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης και άλλα βήματα ή μέτρα που έχουν ήδη προβλεφθεί. Μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας θα ήταν κάτι θετικό γιατί πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι είναι εδώ ο σωστός τόπος για να τα πούμε όλα αυτά και ούτε είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά όπως σας είπα είμαστε υπέρ του να γίνει έκθεση δύο πρωτοβουλία για τα δύο αυτά θέματα που τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά και η ομάδα μου θα υποστηρίξει και τα δύο. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έκαναν τον κόπο να καταθέσουν τροπολογίες και όπως είπα και πριν, ε, ενδεχόμαστε την ένταξη της Λετωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Από τους φιλελευθέρους, ο κύριος Κλίντς είναι ο Σκιώδης, αλλά δεν τον βλέπω. Τον αντικαθιστά κανείς. Από ό,τι φαίνεται όχι. Επόμενη ομάδα. Η πράσινη, ο κύριος Μπρισσέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci, merci Madame la Présidente. Ε, très rapidement, Euh, Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το ανοιχτό πνεύμα που έδειξε. Ε, άρα δεν υπάρχουν σημαντικά πολιτικά προβλήματα. Και στο πνεύμα αυτό άκουσα βεβαίως κύριε Μπάλ την δέσμευσή σα, ε, την οποία επανέλαβαν και οι σοσιαλιστές συνάδελφοι, ότι το θέμα των κριτηρίων σύγκληση ε, και του διεύρυνση ε, δεδομένη της εξέλιξη τη κατάσταση για την οποία έχουμε καταθέσει μια τροπολογία, δεσμεύεστε να συζητηθεί ευρύτατα σε αυτή την, την Επιτροπή. Η προοπτική μιας ε, έκθεσης πρωτοβουλία θα είναι φυσικά ένα πλαίσιο ενδιαφέρον και θετικό. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρχει αυτή η δέσμευση, εμείς αποσύρουμε αυτή την τροπολογία που είναι η 8, καθώς και την τροπολογία 9, εξάλλου που ήταν συγγενική. Αντιθέτως διατηρούμε την συγγνώμη δεν έχω τα γυαλιά μου, 18, που αναφέρεται, ακούσαμε βέβαια τα δικά σε επιχειρήματα, αλλά αναφέρεται στο θέμα της φορολόγησης των επιχειρήσεων και των φόβων που μπορεί να έχουμε από αυτή την άποψη δεν θέλετε να μπει σε αυτό το πλαίσιο, αν και δεν είστε κατά των συμφωνιών επί της αρχής για αυτήν την επιτυχή, αλλά εμείς κατά τη γνώμη μας θα προτιμούσαμε να το σημειώσουμε και αυτή η διάσταση να ενταχθεί μέσα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να το να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον εισηγητή για την εργασία. Ναι, αλλά δεν μας είπατε για την απολογία παριθμών 9 ποια είναι η θέση σας. Ε, ναι, ναι, το είπα. Αλλά μήπως έκανα λάθος το ε, αριθμό. Την αποσύρουμε. Και την 8 και την 9. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Από τους συντηρητικούς, ο κύριος Ζήλε δεν είναι εδώ, ζήτησε ο κύριος Τρέιτσεκ να μιλήσει και τον είναι παρακαλώ. Well, thank you. Thank you, Madam Chair. Uh, the ECRs... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής είναι ο κύριος Ζήλερ, αλλά δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματός του. Δεν θα μιλήσω, αλλά θα διαβάσω τη θέση του πάλι να τονίσω ότι είναι η θέση του κ. Ζήλα και όχι δική μου. Ο σκιώδης εισηγητής ε, του CCR, κ. Ζήλα, ευχαριστεί τον κύριο Πάλτς για την ισορροπημένη και πολύ σημαντική έκθεσή του. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι από τη μια πλευρά δείχνει πως το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει ε, τις ε, την βούληση της Λετωνίας να μπει στην Ευρωζώνη και δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη βυθό ότι οι προσπάθειές της έχουν ε, ε, διαπιστωθεί και ανταμείβονται. Από την άλλη πλευρά το Κοινοβούλιο σαφώς δήλωσε ότι αυτό ακόμα θα πρέπει να γίνει σε σχέση δηλαδή με τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας ε, της επάρκειας σε ενέργεια και της διαφοροποίησης. Αλλά ε, η ανακοίνωση ε, για την εισαγωγή του ευρώ, βελτιώσεις στην εποπτεία των τραπεζών, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των καταθέσεων των ε, αλλοδαπών. Αυτό το πρόβλημα, αυτός ο κατάλογος θα πρέπει να θεωρηθεί από τη λετωνική κυβέρνηση ως ένας κατάλογος εργασιών που δεν θα πρέπει να καθυστερήσει καθόλου εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Αυτά είπε ο κύριος Ζήλαντ. Oh, Συγγνώμη, Πρόεδρο, στο μικρόφωνο μου. Επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε άλλους αγιαγραμμένους ομιλητές. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, αλλιώς ε, εισηγητής. ο κύριο Κάριν, παρακαλώ. Thank ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Εγώ θέλω να σχολιάσω τις 7 συμβιβαστικέ που έχει υποβάλει ο εισηγητής. Νομίζω πως είναι σωστά συνταγμένες και λαμβάνουν σωστά υπόψη το πνεύμα της ε, έκθεσης. Θέλω να τις υποστηρίξω. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κύριε Μπάλτς, θέλετε να πάρετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω νομίζω η συζήτηση μιλάει από μόνη της. Ε, από κοινού, και το τονίζω, από κοινού ε, κάναμε αυτή την προσπάθεια με όλους τους κοιόδης και θέλω πάρα πολύ ε, όλοι μαζί ως Επιτροπή να συστήσουμε στην αδομέλεια να εγκρίνει την ε, ένταξη της Λετωνίας στο ευρώ. Αυτά και στα μετώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, τι τυχερός που είστε. Είναι όλοι εχέφρονοι οι σκιώδει. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Αφού είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα μπορούμε να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Μου δίνετε λίγο μια λίστα ψηφοφορία τη δική μου πολιτική ομάδα για να ξέρω τι ψηφίζω παρακαλώ. Έχουμε λέει και άλλο θέμα στη μερισσία διαταξή. Έτσι μου λέγουν πριν την ψηφοφορία. Τι είναι αυτό? Α, με γενικό προπολογισμό τη Ένωση για το. Εντολή, εντολή. για το οικονομικό έτος 2014 για όλα τα τμήματα. Ε, ο εισηγητή είναι ο κύριο Γκίγκολτ και έχει το λόγο. It seems, ε, that, ε, Από ό,τι φαίνεται, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς όταν θελήσατε να πάτε αμέσως στην ψηφοφορία. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να μιλήσω. ε, για να σοβαρευτώ. Το να δουλεύει κανείς στον προϋπολογισμό είναι δύσκολο όταν δεν υπάρχει πρόταση για τον προϋπολογισμό. Πράγμα που ισχύει σήμερα. Βρισκόμαστε σε αυτή την ηρωνία. Θα προτιμούσα να δουλεύω σε ένα προπολογισμό με αριθμητικά στοιχεία. Αλλά μου λέγει η γραμματεία ότι πρέπει να γράψει την έκθεσή μου έτσι κι αλλιώ και α μην έχουμε προπολογισμό. Οπότε έβαλα μερικές γενικές αρχές ε, που είναι κοντά σε θέσεις παρελθούσες του Κοινοβουλίου, υποθέτοντας ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα από ότι σοφές ε, διαβουλεύσεις στην Κομισιόν για το προϋπολογισμό. Δεν θέλω να τα επαναλάβω τώρα εδώ όλα όσα προτείνω, θέλω μόνο να τονίσω ένα σημείο που μας ε, προκαλεί ανησυχία. Έχουμε δώσει πολλά καθήκοντα νέα ε, στην ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εποπτείας. Τουλάχιστον ε, αυτό το κομμάτι του προπολογισμού μας αναλογεί εμάς. Και ακούω με κάποια αγωνία και έχω θορυβηθεί ότι το καθεστώς που είχαν μέχρι τώρα αλλάζει. Και επειδή ε, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλάζουν ε, οι αρμοδιότητες των οργανισμών ε, των δορυφορικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι επικίνδυνο. για όλους, για τις κοινικέ αξίες, για διάφορες άλλες μορφές και στη φεραγγιότητα, αυτά που λέει ο Μπάλτς, ε, Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που επιφορτίζονται με αυτά τα θέματα και γνωρίζουμε πόσο περίπλοκο είναι. Ταυτόχρονα όμως, δεν έχουμε αντίστοιχη αύξηση ε, των εκάστοτε προϋπολογισμών, είναι περιορισμένη αυτή. Και μάλλον προτιμούν ορισμένα μέλη του Συμβουλίου ένα γενικό κούρεμα. Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν αυτό στον προπολογισμό, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορεί να δίνει περισσότερε και νομοθετικέ αρμοδιότητε ε, σε αυτού του οργανισμού εποπτεία κλπ. Και, και μετά να πούμε ναι, αλλά λεφτά δεν έχουμε. Ε, και έτσι δεν μπορεί να αυξηθεί το προσωπικό σα αναλόγω. Έχω δει την κατάσταση αυτή στο Λονδίνο, όπου Πήγα στα γραφεία της, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και είδα πολλούς νέους ενθουσιώδεις και δυναμικούς που εργάζονται εκεί και δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, αλλά αυτά που πληρώνουν ως μισθούς δεν είναι ανταγωνιστικά στο Λονδίνο και στην ΑΙΟΠΑ το ίδιο περίπου ισχύει, διότι έχουμε νέο ανταγωνισμό από την επόπτη τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι θέμα μεγέθους μόνο, είναι και θέμα του ε, αν πληρώνεις καλούς μισθούς και προσελκύεις τον κόσμο για να είσαι ανταγωνιστικός με τους ε, ε, εθνικούς επόπτες αλλά και με θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, τι θα πρέπει να έχουμε εμείς ως αντικειμενικό σκοπό ότι δεν μπορούμε να νομοθετούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χρηματοπιστωτικά και μετά να μην έχουμε τους πόρους για να δίνουμε την απαραίτητη συνέχεια. Αυτά είναι πάγια αιτήματα της Επιτροπής μας και νομίζω θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα προωθούμε. Για τα υπόλοιπα θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. για να είναι ισόρροπη η έκθεση για τον επόμενο προπολογισμό. Και επίσης κυρία Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να δώσετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πότε θα έρθουν ε, τα αριθμητικά στοιχεία και αν θα δώσουν συνέχεια σε αυτά που ζητεί το Κοινοβούλιο ή σε αυτά που ζητεί η Eurostat και οι τρεις ε, οργανισμοί εποπτείας, η ΕΣΑ. Ή θα βασιστούν στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θέλετε να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τους σκιώδεις ε, εισηγητές ή όχι. Μετά. Ο κύριος Φέρμπερ από το Έλκυνο, πρώτος σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κοιτάξτε, να δούμε τα πράγματα λίγο νυφάλια έχουμε στήσει μια τεράστια μηχανή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω πόσους οργανισμούς έχουμε, 25, 28, 30, κάπου εκεί. Και κάθε επιτροπή αγωνίζεται για το δικό της οργανισμό να γίνει πιο μεγάλος και πιο σημαντικός και εμείς τώρα χτίζουμε κάποιους οργανισμούς που θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητοι. Και δεν διευκολύνει αυτά τα πράγματα, πολλό δε μάλλον που ζούμε καιρούς, μάλλον, πώς να το πω, για την επόμενη επταετή περίοδο θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη φαντασία για να βρούμε περισσότερα χρήματα από ό,τι στο παρελθόν. Λοιπόν, τα πράγματα περιπλέκονται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα απολύτω απαραίτητα και να είμαστε πρόθυμοι να πιάσουμε και το κόκκινο μολύβι και να αρχίζουμε να κόβουμε από αλλού. Εμείς στη δική μας επιτροπή έχουμε αρμοδιότητα για λίγες θέσεις μόνο του προπολογισμού. Και διαρωτώ αν είναι πραγματικά δική μας δουλειά τώρα να υποστηρίζουμε οικονομικά αυτούς που έτσι και αλλιώς στρέφονται εναντίον μας. Τουλάχιστον για μένα δεν με εξέλεξαν γι' αυτό, ούτε για να αυξάνεται η χρηματοδότησή τους. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να τα δούμε με νυφαλιότητα και ηρεμία. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς αυτού δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω αυτό που είπε ο εισηγητής. Το θέμα δεν είναι να διαγωνίζονται οι επιτροπές ποιος έχει το μεγαλύτερο, ωραιότερο και καλύτερο οργανισμό, αλλά αυτό που εμείς πολιτικά επιθυμούμε να μπορεί οργανωτικά να υποστηρίζεται με το απαραίτητο προσωπικό γι' αυτό και τη στελέχωση που χρειάζεται. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Επόμενος ο σκιώδης των σοσιαλιστών, κύριος Γουάγκ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα δέχεστε φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα λεπτό να αρχίζουμε τις εργασίες μας για τη γνωμοδότηση της εικόνας στον προϋπολογισμό, ενώ δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οι δημοσιονομικές προοπτικές 14 με 20 η Επιτροπή Προϋπολογισμών τη συζητάει σήμερα αλλά δεν θα μπορέσουν να αποφανθούν οι συνάδελφοι επίσημα πριν το Σεπτέμβριο. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας αυτή την πολύ λεπτή πολιτική συγκυρία και να γνωρίζουμε ότι δεν είναι βέβαιο το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην προδικάζουμε τι θα γίνει τους τελεπόμενους μήνες. Και γι' αυτό η διατύπωση στην παράγραφο 2 της γνωμοδότησης είναι κατ' εμέ προβληματική γιατί ήδη δέχεται τον προϋπολογισμό του 14 με λιγότερα ποσά, με λιγότερο ύψος. Και στην, ενώ στην παράγραφο 1 ζητούσε έντονα έναν αντικυκλικό προϋπολογισμό. Το κείμενο τελικά θα το πάρουμε αυτή την εβδομάδα και πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον και την αντίδραση της Κομισιόν πριν αποφανθούμε για τις σοσιαλιστικές τροπολογίες. Γιατί ο στόχος ακριβώς στην εικόνα είναι να προεργαστούμε πρώτα να εξετάσουμε λεπτομερώς την πρόταση της Κομισιόν. Το σχέδιο γνωμοδότησης του Σβέν Γκίγκολτ βασίζεται στις πολιτικές προτεραιότητες όπως τη χρηματοδότηση των αρχών επιτήρησης κτλ. Και αυτό είναι σωστό, είναι μια προσπάθεια όμως να παρακάμψουμε το πρόβλημα. Θεμητό αυτό και ενδιαφέρουσες οι προτάσεις της εισηγητή, αλλά και άλλα προγράμματα που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την εικόνα θα μπορούσαν να έχουν την ίδια τύχη, όπως το φυσκαλής. Καταλήγω, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στην εικόνα ακόμα και θα πρέπει να κατατεθούν και άλλες προτάσεις για να ενδυναμωθεί η πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος σκιώδης των φιλελευθέρων, ο κύριος Τόρβαλτζα, αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Είναι κανείς άλλος από τις φιλελεύθερους που θα ήθελε να πάρει τον όχι. Η συντηρητική, ο κύριος Τσίλε, ούτε αυτός είναι εδώ. Μήπως είναι κανείς άλλος συντηρητικός που θα ήθελε να αναλάβει, όχι. Δεν έχω άλλους σκιώδεις από την ΚΟΕ, μήπως κανείς άλλος συνάδελφος θέλει να μιλήσει. Κύριε Λάμπερτ, όχι, αλλά ε, ε, ε, Τότε μπορώ να μιλήσω ως συντηρητικός, μπορώ να μιλήσω ως γκουε, Α, όχι, όχι. Εννοούσα άλλους, όχι να εκπροσωπούν σκιώδεις. Η τριτοκλασάτη εννοούσα. Που, σχεδόν ποτέ δεν παίρνουν το λόγο. Λοιπόν, κύριε Γκίγκουλ, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Συμφωνούν όμως να σας απαντήσουν κραπτός. Ορίστε έχετε το λόγο. Καλά, στα γερμανικά. Εάν απουσιάζουν δεν μπορούν να μας απαντήσουν. Λογικό μου ακούγεται. Αν κατάλαβα καλά όμως, τέλη του μηνός Επιτέλους αρθούν έρθουν και τα ποσά. Ε, μεθαύριο είναι περίπου το τέλος του μηνός. Κάποια στιγμή ελπίζω να μας έρθουν και τα στοιχεία. Κυριακή κοντή γιορτή. Ε, περιμένω και τις τροπολογίες των συναδέλφων. Μήπως μάθω και που χρηματοδοτούμε αυτούς που στρέφονται εναντίον μας. Όπως ακούσαμε. Τουλάχιστον αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το εξής. Το έφρακ θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται που είναι η μεγαλύτερη επιδότηση που δίνουμε εδώ πέρα και αν είναι ξεχωριστή διαδικασία, ε, είναι ένα θέμα που απασχολεί την έκθεση του κυρίου Στόλογιαν. Ε, από εκεί και πέρα να πω στο Λίαμνο ε, μόνο ότι το σημείο 2 δεν πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι έτσι. Δεν λέω πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι το υπόλοιπο του κοινοτικού προϋπολογισμού, αυτό που λέω είναι όταν κάνεις πάντα δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να μιλάς και για οικονομίες και να σκέφτεσαι ε, και που θα περικόπτεις. Αλλά στην Επιτροπή Οικονομικών δεν θα πρέπει να κάνουμε περικοπές στις επενδύσεις του μέλλοντος. Θυμάμαι στην πρώτη συζήτηση που κάναμε για την έκθεση μου, αυτό ακριβώς είπες. Και θεωρούσα ότι όλα αυτά πηγαίνουν σε δική σου κατεύθυνση. Ας πούμε δεν μπήκα στο γεωργικό προϋπολογισμό, είχα την ευγενή καλοσύνη να το κάνω αυτό, παρόλο ε, που είχαμε διαφωνήσει τότε λίγο με τη δική σου θέση. Ε, δεν έχω πρόβλημα να σκεφτώ που μπορούμε να κάνουμε οικονομίες και θα σας επαναλάβω την πρόταση των πρασίνων. Τα χρήματα, ας πούμε, ε, που επενδύουμε για υλικό δημοσίων σχέσεων, ακόμα και αν είναι για το ευρώ, δεν θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλα τα ποσά. Δεν ξέρω, μπορεί αυτή τη φορά να με παρακολουθήσετε, αλλά δεν έχουμε εμείς πολλούς τομείς όπου μπορεί να πέσει γερό μαχαίρι. Ε, ε, αυτά στον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι αλλού ε, σε άλλες επιτροπές για να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις του μέλλοντος και να κόψουμε εκεί που χρηματοδοτούμε εδώ. Πρέπει να πάμε να ψαρέψουμε λοιπόν σε άλλα νερά. Ευχαριστώ. Χρονοδιάγραμμα η Πρόεδρος. Αυτή ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών προβλέπεται για τις 18 Ιουλίου. 5 Σεπτεμβρίου συζήτηση των τροπολογιών και βάσει του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής Προπολογισμών κανονικά θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου επίσης. Ορίστε. Ο κύριος Κοζές, κυρία Πρόεδρε. Το είπε προηγουμένως ο συνάδελφος των σοσιαλιστών, αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς πώς θα δεσμευτούμε, πώς θα γνωμοδοτήσουμε, δεν ξέρουμε το γενικότερο προέσιο και λυπούμε για την απουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλά θα το δούμε αυτό, ε, μέχρι τότε θα ξέρουμε. Μα δεν έχει νόημα τώρα να ε, ε, ορίζουμε έτσι τα χρονοδιαγράμματα και μετά να τα αναβάλουμε. Είναι προσφυλές μας άθλημα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και θα πρέπει από την αρχή να προσανατολιζόμαστε σε μειώσεις, σε περικοπές και να μην κάνουμε τη δουλειά μας σωστά γιατί δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους. Για πράγματα που εμείς εσπίζουμε. Έχετε δίκιο κύριε Κοζές, αλλά ε, η γραμματεία της Επιτροπής μας εδώ ε, κάνει κάποιες ενδεικτικές προβλέψεις. Δεν σημαίνει τίποτα. Ενδεικτικά είναι οι ημερομηνίες. Ναι, κυρία Πρόεδρε, είδαμε τα ενδεικτικά. Όπως έλεγε ο Πιέρ Ντάκ, ο Γάλλος κομικός, ότι είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το μέλλον. Να πω κάτι εγώ, γι' αυτό λέει ο κύριος Γκίγολτ. Ναι, και εγώ το βρίσκω πολύ περίεργο. Να γράφουμε εκθέσεις ε, χωρίς να έχουμε την ουσία του θέματος και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον Ζαν Πολ θα πρέπει να το λύσουν αυτό οι συντονιστέ. Πώ γράφει κανεί έκθεση χωρί να έχει την πρόταση για τι γραμμέ του προπολογισμού με τα αντίστοιχα ποσά. Είναι σπάνιο αυτό και μυστήριο. Και ο Καλ Βάλεντιν, ο Γερμανό ε, είχε πει και αυτό ότι οι προβλέψεις είναι δύσκολε, ιδίω όταν αφορούν το μέλλον. Λοιπόν, τι είναι όλο αυτό το εγχείρημα, τι νόημα έχει να μου το εξηγήσετε, αλλά εγώ επειδή είμαι φαντάρο εδώ ταγμένο, κάνω ό,τι μου λένε. Κοιτάξτε, και εγώ θα αναρωτιόμουν γιατί συζητάμε τον προϋπολογισμό του 2014 ήδη, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών πρέπει να εξετάσει τη γνωμοδότησή μας. Χρειάζεται ένα χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Το σημαντικό είναι η διορία κατάθεση των τροπολογιών που λήγει 18 Ιουλίου. Και μετά θα δούμε. Η ψηφοφορία για τις 5 παρα 20 προβλέπεται, δεν έχουν έρθει όλοι ακόμα, γι' αυτό διάλειμμα μέχρι τότε στις 5 παρα 20 ακριβώς για να ψηφίσουμε. Και μετά φαίνεται ότι η κυρία Μπόλτ θα εμφανιστεί για να προεδρεύσει μετά την ψηφοφορία. Αλλιώς θα συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, διάλειμμα. Steht auch in der Tagesordnung. Το λέει και η ημερήσια διάταξη, άμα δεν το είδες. Είστε έτοιμοι, τότε σας ευχαριστώ. Πρώτα δοκιμή. Μήπως κανείς δεν έχει την κάρτα του και εγώ δυστυχώς δεν έχω την κάρτα μου. Άλλος, άλλος, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Άρχισε, έληξε, εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Μάλιστα, ικανοποιήθηκαν 22. Μάλιστα. Παράγραφος 1, αρχικό κείμενο, περ, τα, χες, εγκρίνεται. Δυο παράγραφος υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Τροπολογία δύο υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Η 5α έχει αποσυρθεί. Συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Για να δούμε πού είναι η συμβαστική ε. Ναι, ε, συμβιβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβιβαστική σιγματάφη υπέρ κατά αποχές. Προφορική τροπολογία στην συμβιβαστική ζήτα. Εγώ είμαι κατά. Α, είναι κανείς άλλος κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ωραία, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε λοιπόν. Θα μπορούσαμε και απλώς να την είχαμε καταψηφίσει, αλλά τέλος πάντων. Συμβαστική ζήτα, όσοι είχε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία των πρασίνων επί της 18 Θα τη δεχτούμε την προφορική. Δεν έχει κανείς αντίρρηση λοιπόν. Αν υπερψηφιστεί θα καταπέσει η αρχική. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Επαλήθευσης. κάνουν οι μου εκεί κάτω. Λοιπόν, ένα ακόμα ψήφο στους κατά. Λοιπόν, απορρίπτεται όντω και τώρα η αρχική 18 υπέρ κατά ίσως να επαληθεύσουμε γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Η αρχική τροπολογία 18 η αρχική. Ακόμη 5 έληξε απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 20 υπέρ κατά χες εγκρίνεται σε δύο τμήματα για την 22. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε όλα τις αιτιολογικές να τις κάνουμε μαζί μέχρι το τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ηλεκτρονικό στο σύνολο ένας ακόμη εντάξει 35 μαζί με μένα υπέρ κάποιος άλλος κατά και δύο αποχές ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον Μπούρκχαρτ Τώρα ακόμη ένα διαλυματάκι μέχρι να έρθει ο Υπουργός ή η Υπουργός στις 5. Δεκάλεπτο διάλειμμα. Okay, so, uh, I... Λοιπόν, χαιρετίζω τον Υπουργό προεδρεύοντα του Συμβουλίου Μάικελ Νούναν που έρχεται για τον συνήθι διάλογο στα τέλη της Προεδρίας και μάλλον θα είναι ικανοποιημένοι για πολλά επιτεύγματα τους. Εγώ τουλάχιστον είμαι. Θα ακολουθήσουμε τον συνήθι τύπο 10 λεπτά για τον Υπουργό και μετά 5 λεπτές ερωταπαντήσεις και σας παρακαλώ εκ των προτέρων αν είστε σύντομοι και κάνετε ερωτήσεις και όχι δηλώσεις τότε μπορεί να υπάρξει χρόνος και για τη συνέχεια πράγμα το οποίο είναι συνήθως πιο ενδιαφέρον. Ορίστε Μιχαήλ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ήμουν εδώ τον Ιανουάριο και είμαι ευτυχής που βρίσκομαι και πάλι όπεν αυτή τη Επιτροπής στα τέλη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Είχαμε πέντε επίσημα Συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ και ένα άρτυπο την περασμένη εβδομάδα στο Δουβλίνο. Ελπίζω πως και την επόμενη εβδομάδα θα έρθω γιατί έχουμε άλλη μια άτυπη ε, σύσκεψη στο Συμβουλίο για να δούμε αν θα μπορέσουμε να συμβολήσουμε ε, στο Συμβούλιο για την ε, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πριν ξεκινήσει ακριβώς η Προεδρία μας, ε, εμεί δαπανίσαμε πολύ χρόνο σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να γνωριστούμε μεταξύ μας και έχουμε συνεργαστεί μαζί σας ως συνομοθέτες για διάφορα θέματα διάφορους φακέλους και πιστεύω πως αυτό το κάναμε με θετικό και επικοδομητικό τρόπο. Επιτύχαμε πολλά από αυτά που είχαμε αρχικά ορίσει ως στόχο τον Ιανουάριο και Πρόκειται για προδιαγραφές και για φιλάδοξες δέσμες προτάσεων. Είχαμε σχεδιάσει να ασχοληθούμε με την οικονομική διακυβέρνηση βασικά μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και να συμφωνήσουμε για το διπλό πακέτο για την οικονομική εποπτεία της Ευρωζώνης, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Μιλήσαμε ε, και πάλι και επίσης στοχεύσαμε συμφωνία για τις κεφαλιακές ε, απαιτήσεις και για την ε, ανάκτηση ή διάλυση τραπεζών. Εμείς συμφωνήσαμε για τα MIFID, για το μάρα και για την οδηγία περιπιστώσεων. Ενώ αρχικά υπήρχε συμφωνία στο πρώτο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, μπόρεσαν τα κράτη-μέλη που ήθελαν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της εισαγωγής του φόρου για επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σημαντικές ενδείξεις για το επίπεδο της αμεροληψίας της δικής μας Προεδρίας, καθώς διευκολύναμε άλλους να ξεκινήσουν εργασίες για ένα κείμενο που εμείς δεν σκοπεύαμε να συνυπογράψουμε. Είχαμε και διάφορες άλλες προτεραιότητες σε φορολογίες που σκοπεύαμε να προωθήσουμε τις συζητήσεις για τις ε, ε, ε, κοινές ε, ε, κοινή φορολόγηση των ε, εταιριών, να υιοθετήσουμε το πρόγραμμα Φισκάλης, να δουλέψουμε κατά των, ε, της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης, για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τον ετήσιο προπολογισμό, μπορέσαμε να το διεκπαιρεώσουμε αποτελεσματικά όσον αφορά τον ετήσιο προπολογισμό του 2013 και την προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών για το 2014. Σημαντική πρόοδος δε διατεύχθη στην ατζέντα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γιατί ήταν πολύ σημαντικό να γίνουν βήματα για την νομοθεσία όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και κάναμε επίσης σημαντική πρόοδο στην πρόθεση αυτής της ατζέντα αυτών των θεμάτων που ήταν σημαντική όχι μόνο για την Ελλανδική Προεδρία, για ολόκληρη την Ένωση. Όπως επίσης ε, επιτύχαμε πρόοδο στην ε, οδηγία περί κεφαλαικών απαιτήσεων που θα βελτιώσει το τραπεζικό σύστημα. Ε, συμφωνία επί του εποπτικού μηχανισμού και τροπολογίες για την ε, σχετική νομοθεσία ώστε να βελτιωθεί ο τραπεζική, η τραπεζική εποπτεία σε ολόκληρη την Ένωση. Έγιναν δύσκολε συζητήσει όσον αφορά την ανάκτηση ή την διάλυση τραπεζών ε, και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο ο φάκελο και αυτό στον τομέα τη συνεργασία με τον ε, Κοινοβούλιο για αυτό το σημαντικό φάκελο. Φυσικά μένουν και άλλα να γίνουν, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόγραμμα εγγύησεων για τι καταθέσει. Ωστόσο, η συμφωνία για την ε, ανάκτηση ή την διάλυση τραπεζών είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση πριν προχωρήσουμε στο σχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων. Και αυτό είναι καλά κατανοητό σε ολόκληρη την ενόηση. Ως Προεδρία, ωστόσο, γνωρίζουμε και προσέχουμε και άλλα θέματα της ε, ε, της χρηματοπιστωτικής ε, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ελπίζουμε πως οι σχετικές οδηγίες θα ολοκληρωθούν σε πρώτη ανάγνωση στον επόμενο μήνα. Επίσης έγιναν βελτιώσεις στην οδηγία περί διαφάνειας που θα αυξήσουν την ελκυστικότητα των... της αγοράς για τους μικρομεσαίους. Και τέλος την τελευταία, την περασμένη Παρασκευή κάναμε ε, συμφωνία για τη ΜΥΦΙΤ και ΜΥΦΑ, οπότε πιστεύω πως θα προχωρήσουμε και σε επικοδομητικό τριμερή διάλογο για αυτούς τους πολύ σημαντικούς φακέλους. Για τα θέματα της αγοράς συμφωνήσαμε για το ΜΑΡ τις τελευταίες μέρες είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία όσον αφορά τα επενδυτικά προϊόντα λιανικών ε, πωλήσεων, το TRIP, και έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για την τέταρτη οδηγία περί νομιμοποίησης παρανόμων προσόδων. Σημαντική πρόοδο έχουμε κάνει και στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Έχουμε φτάσει σε συμφωνία στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Εκεί όπου δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσαμε δε τις ε, συζητήσεις, ε, τις έχουμε προετοιμάσει για να τις παραδώσουμε στην επόμενη Προεδρία ώστε να ολοκληρωθεί και η συμφωνία. Είναι σημαντική συνεργασία μεταξύ των Προεδριών ώστε να διατηρηθεί η όθηση τη εργασία του Συμβουλίου Συμβουλίου. Εμείς συνεργαστήκαμε αγαστά με τους συναδέλφους της Κύπρου και με τους συναδέλφους της Λιθουανίας. Υπάρχει περισσότερη δουλειά βέβαια για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Σημαντική ατζέντα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με 16 νομοθετικές ε, προτάσεις και νέες προτάσεις που δημοσιεύονται κάθε μήνα. Οι συζητήσει, γίνονται στο Κοινοβούλιο, θέλουμε να βελτιωθούν όντω οι νομοθετικές αυτές προτάσεις και από αυτό, γι' αυτό αντλούμε από την εμπειρογνωμοσύνη των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Βασικό μα στόχο πρέπει να είναι η σύνταξη νομοθεσιών υψηλού επίπεδου που θα μας επιτρέψουν γρήγορα να μπορέσουμε να έχουμε τα επιθεμητά αποτελέσματα. Είναι μια λογική προσέγγιση πιστεύω και μας έχει εξυπηρετήσει. Τα διδάγματα που αποκαμίσαμε από τι πρόσφατες κρίσεις ε, την οικονομική και την χρηματοπιστωτική ε, οδήγησαν σε αναθεώρηση πολλών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων ε, αλλαγές στις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές, εισαγωγή τραπεζικού και υποπτίας, μεγαλύτερη εστίαση στα χρέη, ε, μνημόνια, πακέτα δημοσιονομικά πακέτα για τα διάφορα κράτη, ε, τα κράτη-μέλη κρίνονται για το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στους μεσοπρόθεσμους στόχους τους, ε, έγκαιρη προειδοποίηση για την διαδικασία υπερβολικού χρέους. Υπάρχει παρακολούθηση ελλείμματος, υπάρχει Επίσης ε, παρακολούθηση και υποπτία των τραπεζών. Θέλουμε να έχουμε συμφωνία για το διπλό πακέτο, η υποπτία για τα κράτη με μεγάλα χρέη ελλείμματα <clears throat> θα πρέπει να επιταχυνθεί. Το διπλό πακέτο έχει αρχίσει να ισχύει από τον Μάιο. Και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμένου είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση του ότι τα κράτη-μέλη θα συζητούν τα δημοσιονομικά τους προγράμματα με τους εταίρους τους της Ένωσης δύο φορές το χρόνο να συστήνεται ένας οδικός χάρτης έτσι ώστε η λειτουργία να είναι πιο ομαλή και πιστεύω πως έχουμε επιτυχία αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και θα διευκολύνουμε και τη διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμένου ώστε να ολοκληρωθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα. Αν και δεν είναι συγκεκριμένα θέμα οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αναφερθώ στην πολυμερή δημοσιονομική αρρωγή προς την Γεωργία και άλλα κράτη, όπου αυτός ο φάκελος δεν είχε προχωρήσει εδώ και κάποιο χρόνο και είμαι ευτυχής που μπορέσαμε να βρούμε μια κατάλληλη λύση. Επιτύχαμε περισσότερα στη φορολογία από ό,τι περιμέναμε. Ήδη αναφέρθηκα στη συμφωνία στο ΕΚΟΦΗΝ που επιτρέπει σε διάφορα κράτη-μέλη να εισάγουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η Προεδρία ήταν ε, δραστήρια και προώθησε διάφορα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής ο Επίτροπος ΕΜΕΤΑ και όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι έτοιμοι να αγωνιστούν κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης. Έχουν ήδη συμφωνήσει από τον Απρίλιο και επί της εντολής για να μπορέσει η Κομισιόν να ξεκινήσει συζητήσεις και με τρίτες χώρες όσον αφορά την φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Είχε υπάρξει συμφωνία όσον αφορά το FiscalNet που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της απάτης. Αναμένεται βέβαια η έγκριση του προπολογισμού. Επίσης έχουμε συμφωνήσει για την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης. Έχουμε προβλέψει και τον μηχανισμό αντιστροφής του βάρους απόδειξης ε, όσον αφορά την φοροδιαφυγή, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα ε, έσοδα στις οικονομίες των χωρών μας και υπό την, κώδικα, υπό τον ομάδα του κώδικα διοντολογίας έχει υπάρξει συμφωνία ε, στο Συμβούλιο ε, του Ιουνίου. Δεν μπορέσαμε όμως να έχουμε συμφωνία όσον αφορά την οδηγία περί φορολόγησης ενέργειας. Ε, έχουμε όμως μιλήσει για ένα ελάχιστα επίπεδα τελών για τα ενεργικά προϊόντα και για κάποιες εξαιρέξεις στην εξάμενη αυτή περίοδο που ήταν πολύ σύντομη θεωρούμε πως ε, προήγαμε την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα συνολικό πιστωτικό σύστημα ώστε οι τράπεζες μας να αρχίσουν και πάλι να δανείζουν στις επιχειρήσεις μας. Οι συνθήκες είναι πολύ βασικές αλλά όχι επαρκείς για να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο δραστήρια, πιο θαραλέα, ώστε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια στρατηγική ενδυνάμωση της οικονομίας ε, καθώς ε, οι τράπεζες έχουν πάψει να δανείζουν μετά από την μόχλευση, μετά την κρίση και γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δουν πώς ε, θα λειτουργήσουν σε συνεργασία ώστε να διοχετευθούν οι διαθέσιμες αποταμιεύσεις προς τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες. Το πρόσφατο πράσινο βιβλίο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι σημαντική εξέλιξη και δείχνει ότι είναι μια πολιτική κλειδί για την Ευρώπη. Ήμασταν δε δραστήριοι όσον αφορά την προώθηση της ατζέντα για την ανάπτυξη, αλλά ε, προβλέπεται Μάλλον η συζήτηση σχετική από στο ΕΚΟΦΗΝ ε, οδήγησε στην απόφαση της δημιουργίας μιας ομάδας ψηλού επίπεδου για την χρηματοδότηση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ε, ε, ενισχύσαμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ώστε και να βοηθήσει και αυτή στη σταθεροποίηση των κρατών μελών. Πολλά δεν έγιναν όσον αφορά τη λογιστική, την οικονομικό συντονισμό καθώς και την νομοθεσία περί του τραπεζικού συστήματος. Περισσότερα βέβαια θα πρέπει να γίνουν και θα ήθελα να έχω τη στήριξή σας και για την επόμενη Προεδρία, ιδιαίτερα όσον αφορά την έγκριση της νομοθεσίας περί τραπεζικής ένωσης. Ο ρόλος του νομοθέτη είναι να διευκολύνει τη συμφωνία και με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο φυσικά καμία Προεδρία δεν μπορεί να επιβάλλει ε, λύσεις. Ως Προεδρία είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε συγκρούσεις συμφερόντων, απόψεων και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε λύσεις που να βρίσκουν σύμφωνο στους περισσότερους. Μπορεί να μην συμφωνούσαμε πάντοτε το περασμένο εξάμεινο, αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να υπάρξει συνένεση σε δύσκολα ζητήματα και τελικά η συνεργασία όλων μας είναι σημαντική για να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα για τους ε, ψηφοφόρους μας. Θεωρώ πως έχουμε πάει καλά μετά από έξι μήνες και σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. εντυπωσιακό ο κατάλογος των θεμάτων που καταφέρατε να προωθήσετε. Ε, κληρονομήσατε πολλά ε, και αποτελματωμένα ζητήματα. Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την απογοήτευσή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ε, αλλά τονίζουμε πάντα ότι δεν φταίει η Ιρλανδική Προεδρία αυτή καθ' αυτή. Γενικότερα, εμείς εργαζόμαστε πιο γρήγορα η σειρά ετών από ότι το Συμβούλιο. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις πεντάλεπτες ερωτήσεις και απαντήσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρώτος ο Ζαν Πολ Γκοζές, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύον. Δεν αμφιβάλλω. Ούτε στιγμή δεν αμφιβάλλω για την προσωπική σας προσήλωση και για τη σημαντική δική σας ε, εργασία. Κοιτάξτε τώρα που σας επενώ, αν δεν έχετε τα ακουστικά σας, θα ακούσετε μόνο τις κριτικές. Οπότε προτιμώ να επαναλάβω. Ε, πρόεδρε, έλεγα ότι δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι είστε προσωπικά πολύ ε, προσιλωμένος και έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να προωθήσετε τα διάφορα θέματα. Οπότε από αυτή την άποψη μπορείτε να πείτε όντως ότι η Ελλαδική Προεδρία εργάστηκε επιμελώς. Επιτρέψτε μου όμως να δω τα πράγματα όπως οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, γιατί αυτούς εκπροσωπούμε εμείς εδώ. Και για τους συμπολίτες μας η Ευρώπη δεν προχωρεί, δεν προχωρεί. Τα εκλογικά αποτελέσματα Κυριακή ρε Κυριακή, όλες οι αρνητικές ε, εξελίξεις και ε, ομιλίες δείχνουν στις χώρες ότι ούτε εσείς ούτε εμείς καταφέραμε ε, να κάνουμε στους πολίτες να καταλάβουν και να εκτιμήσουν τη δουλειά μας. Γιατί πρώτον τα σημαντικά θέματα είναι σε εμπλοκή, μόλις θύμισε ε, την πρόταση που ψηφίσαμε η Πρόεδρος, γιατί είναι σπάνιο ε, πράγμα να αμφισβητεί κανείς το σύνολο του Συμβουλίου, όχι την Ιρλανδική Προεδρία και την αδυναμία των κυβερνώντων, ε, ακόμα και αυτών που είναι από την ίδια πολιτική παράταξη, να βρίσκουν κοινέ λύσεις απέναντι στα θέματα που τους απασχολούν. Το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, εμείς εργαστήκαμε γρήγορα και μάλιστα όχι άσχημα θα έλεγα. Και με τη συνένεση που δείχνει ότι μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις. Δυσκολευόμαστε να τα εξηγήσουμε αυτά και να τα καταλάβουν οι πολίτες. Επίσης δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ότι δεν έχει τελειώσει η κρίση. Και δεν σας βοηθούν ε, οι ομολογοί σας γιατί το γυρνούν στις χώρες τους. Ε, λέγουν ότι αλλού έχουν προβλήματα, όχι οι ίδιοι, γιατί θα έχουν λύσει. Καθόλου δεν τα έχουν λύσει. Και αυτό που επιθυμούμε από μια προεδρία, εσείς με μεγάλο ε, σθένος και θάρρος και παρησία προσπαθήσατε να το κάνετε, να ευθυγραμμίσουμε τις χώρες. Και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώνουμε ότι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που χαρακτηρίζονται από ορισμένου και μέχρι ζωτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε εμπλοκή. Εγώ κατανοώ τα εθνικά συμφέροντα, κάθε χώρα τα συμφέροντά τη υπερασπίζεται. Αλλά νομίζω ότι οι συμπολίτε μα περιμένουν άλλα από την Ευρώπη. Και μάλιστα όσοι είναι ευρωπαϊστές ανησυχούν γιατί βλέπουν αδιαφορία, περιφρόνηση ακόμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω κάποιων ατυχών δηλώσεων του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μάλλον δεν ε, ήλεγχε αυτά που έλεγε αρκετά. Δεν θέλω καθόλου να σας ψέξω για τη δική σας εργασία, αλλά ε, σίγουρα θα διαβάσατε την πρόταση που ψηφίσαμε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να μου απαντήσετε τι φρονείτε από αυτής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζέσου όλοι γνωρίζουμε σε όλες τις χώρες μέλη την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές όχι μόνο στη δική μας χώρα και στην Πορτογαλία και αλλού. Πληρώνουμε ακριβά για τις αμαρτίες του παρελθόντος και η δημοσιονομική διόρθωση δεν είναι ποτέ κάτι εύκολο αν περικόπτονται οι δαπάνες, αυτό έχει επιπτώσει τις υπηρεσίες και αν αυξάνονται οι φόροι, αυτό επηρεάζει τα εισοδήματα πολλών. Και φυσικά η ανεργία σε τέτοιες περιπτώσεις πάντοτε αυξάνεται. Γι' αυτό η Ιρλανδική Προεδρία επέλεξε τη σταθερότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη ως τα κύρια θέματα της. Γιατί η διόρθωση των ελλημάτων και η βιωσιμότητα του χρέους είναι μεν απαραίτητα μέτρα αλλά δεν καταλήγουν μακροπρόθεσμα να πετύχουν τους στόχους που έχουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε ως ολόκληρη την Ένωση να κάνουμε τις δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται και γνωρίζουμε τη συζήτηση που γίνεται σε όλες τις χώρες για τα προγράμματα λιτότητας, για τα διορθωτικά προγράμματα, αν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Εμείς ως Προεδρία θεωρήσαμε ότι το θέμα δεν ήταν να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα αντί άλλου, αλλά μαζί. Αυτό πρέπει να επεξεργαστούμε. Ως προς το τι θα θέλαμε να γίνει και τι ζητούσαμε να γίνει ως Προεδρία, εμείς θεωρούμε ότι τα διορθωτικά προγράμματα μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν, αλλά ότι υπάρχει πολύ λίγη πρόοδος που σημειώνεται για τη συμπλήρωση της αγοράς και όμως αυτό επηρεάζει το ΑΕΠ όλων των χωρών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί 180 δισεκατομμύρια περίπου το χρόνο σε επενδύσεις και αυτό που καθυστερεί τα πράγματα είναι η χρηματοδότηση τους βέβαια από τρίτα μέρη. Το αμερικανικό πρότυπο λέει ότι 75% της χρηματοδότησης για τη βιομηχανία προέρχεται από πηγές εκτός των τραπεζών. Νομίζω ότι εμείς εξαρτώμεθα υπερβολικά από τις τράπεζες στην Ένωση, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό στην άτυπη συνάντηση του Δουβλίνου ε, υπάρχει ένα, μια πράσινη βίβλος που θα μιλάει για τις εναλλακτικέ λύσεις προς την τραπεζική χρηματοδότηση. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα ότι δεν μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα σε έξι μήνες αλλά τουλάχιστον τα απαραίτητα. Ευχαριστώ. για τους σοσιαλιστούς ο Λίαμ. Ευχαριστώ Σάρων. Κύριε Υπουργέ, επιμείνατε ότι υπήρξαν πρόοδοι στην οικονομική διακυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα ή έλλειμμα δημοκρατίας και το είδαμε πρόσφατα και όταν η Κομισιόν καθόρισε στόχους μείωσης των ρημάτων πολύ πιο περιοριστικούς και γρήγορους από ό,τι προτείνει, πρότεινε η εξάμετρος και η δίμετρος. Και νομίζω ότι με περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο θα μπορούσαν να αποφευχθεί λάθη και δεν θα αναγκαζόταν η Κομισιόν να αναθεωρήσει πάλι τις προβλέψεις της για πολλές χώρες της Ένωσης όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ισπανία κλπ. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Ράσμουσεν σήμερα. Είναι μέλος του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είπε ότι στην προσεχή φάση της Οικονομικής Ένωσης θα χρειαστεί ένα, μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση ελεγχόμενη από τις δημοκρατικές, από τα δημοκρατικά κέντρα. Αυτά περίπου έλεγε το Κοινοβούλιο και στην έκθεση Τάισεν, δηλαδή ότι σε κάθε επίπεδο λήψη αποφάσεων πρέπει να υπάρχει ένα δημοκρατικό αντίβαρο. Ενώ ο κύριο Άσμουσεν μα λέει ότι μπροστά στο ε, Ευρωζώνη και το Συμβούλιο πρέπει να ενδυναμωθούν οι δικαιοδοσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα πολύ περισσότερο να κάνει τον έλεγχο το Κοινοβούλιο από ότι μια επιτροπή από εθνικά. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού. Αν θα μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στους ε, Λιθουανούς που θα αναλάβουν την Προεδρία μετά από εσάς. Well, Για το θέμα της διακυβέρνησης. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, δεν εφαρμοζόταν με δίκαιο ακριβώς τρόπο. Νομίζω ότι ε, το διορθώσαμε και οι συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βοηθούν πολύ. Γίνεται μεγάλη διαβούλευση με τις ε, χώρες τις ενδιαφερόμενες φορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφερε στο Συμβούλιο προς έγκριση την πρότασή της και η οποία πρόταση εγκρίθηκε χωρίς τροπολογίες. Βεβαίω, σε κάποιε χώρε δόθηκε επιπλέον χρόνο για να κάνουν τι απαραίτητε προσαρμογέ του, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα επιχειρήματα και να ακούμε τα όσα λέγονται για την έλλειψη ζήτησης, για την έλλειψη καταναλωτικής ζήτησης ε, στην αγορά και χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο κάποιες ε, οικονομίες και αυτό μου φαίνεται λογική προσέγγιση. Προχωρούμε προς τη Δημοσιονομική Ένωση, παραμένουν οι ίδιοι οι κανόνες, δεν έχουμε αποστεί, αλλά ελήφθη μια απόφαση να δοθεί κάποια ευχέρεια σε κάποιες χώρες χρονική για να προσαρμοστούμε τους κανόνες για τη ε, Δημοσιονομική Ένωση. Και αυτό μου φάνηκε εξόχως ε, λογικό και ευθυγραμμισμένο με την καλύτερη μακροοικονομική σκέψη. Ε, τώρα, αν ήταν καλύτερες αποφάσεις, αν υπήρχε μια επιτροπή του Κοινοβουλίου που θα συμμετείχε στη διαδικασία ή όχι, ομολογώ ότι δεν ε, το γνωρίζω. Γενικά είμαι πάντα υπέρ του εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρετε ότι είναι η τρίτη μου προεδρία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ε, και το Κοινοβούλιο έχει και περισσότερα πλεονεκτήματα και ε, εξουσίες ε, ως συνομοθέτης και μέχρι τα τέλη του μηνός θα έχουμε 10 ίσως και 11 θέματα από τα οποία 7 είναι σε πλήρη συνομοθετική διαδικασία με το Κοινοβούλιο. Άρα θεωρούμε την Προεδρία μας ως πολύ επιτυχή. Αλλά η Ευρώπη είναι συνεχώς υποδιαμόρφωση. είναι ένα εγχείρημα το οποίο συνεχώς ε, εξελίσσεται. Διάβαζα τη βιογραφία του Τόμας Τζέφερσον και τις συγκρούσεις που είχε με τον Άντρου Χάμιλτον στη δεκαετία του 1780-1790 μέχρι το τέλη του αιώνα. Και αντίστοιχα με αυτά που συμβαίνουν τώρα ε, στην Ευρώπη έγιναν και στην Αμερική και πόσο κοντά ε, ήταν ε, οι αποφάσεις και τι επηρέασε τις αποφάσεις και πόσο μικρά ήταν τα περιθώρια. Και αν είχαν αποφασίσει κάτι διαφορετικό θα ήταν σε πολύ διαφορετική εξέλιξη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, η Ευρώπη δεν είναι κάτι το στατικό, είναι δυναμική εξέλιξη ανάλογα με το χρόνο που περνά. Και μπορεί να γίνονται μεγάλα άλματα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη και αυτό πάντα είναι απάντηση ως έναν καταλήτη από τη, ε, τραπεζική ε, για να γίνει τραπεζική ένωση και δημοσιονομική ένωση χρειάστηκε ως καταλήτης η οικονομική καταστροφή και η κρίση. Τώρα μπορεί κάποιος άλλος καταλήτης να μας κάνει να προχωρήσουμε με άλματα. Η Ευρώπη δεν προχωράει ποτέ με βηματάκια, άλματα κάνει πάντα. Uh, από τους φιλελευθέρους ο Φίλιπ Ντεμπάκερ στα αγγλικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Προεδρία για το περασμένο εξάμεινο και τη δουλειά που προσπαθείτε να κάνετε ως διαμεσολαβητές όχι μόνο σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα και χρηματοπιστωτικά, αλλά και σε άλλα που έχουμε δει ότι έχουν οδηγηθεί σε εμπλοκή σε άλλες επιτροπές. Αυτά από πλευρά μου. Ίσως δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Το πρώτο μπορεί να σας φανεί λίγο φιλοσοφικό τις τελευταίες δύο ημέρες ακούσαμε διάφορες δηλώσεις από τις Ηνωμένε Πολιτείε, τον κύριο Μπερνάνκη πρώτο και οι αγορές ε, αντέδρασαν πολύ βαριά και αρνητικά. Μετά από δύο μέρες ε, είδαμε τα ίδια από την κινέζικη πλευρά με μια δήλωση που έλεγε ότι θα υπάρξουν και κάποια προβλήματα και στο δικό τους χρηματοπιστωτικό σύστημα και επίσης γνωρίζουμε ότι τελικά δεν συνδέονται μόνο οι χώρες μας μεταξύ τους ε, δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά, είναι παγκόσμιο αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως βλέπουμε ότι δεν καταφέρνει να συμφωνήσει το Συμβούλιο για σημαντικά θέματα όπως είναι η Τραπεζική Ένωση, αλλά και ε, την εκαθάριση τραπεζών. Αλλά βλέπουμε ότι είναι μεγάλη αστάθεια και αβεβαιότητα παγκοσμίω και από την Αμερική και από την Κίνα και γενικότερα. Εσείς Πώς βλέπετε να προχωρούν αυτά τα θέματα, μήπως είμαστε υπερβολικά αργοί και με συγκεκριμένα αποτελέσματα και πάλι κατακαιρματίζεται η αγορά, η χρηματαγορά στην Ευρώπη. Το είπατε κι εσείς, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμποδίζονται στη χρηματοδότησή τους και έχουν προβλήματα ρευστότητας. Λοιπόν, υπάρχουν κανένα δύο θέματα, οι προτάσεις που θέλετε να έρθουν ε, σύντομα τις επόμενες εβδομάδες ή και μήνες για να βοηθηθούν οι εταιρείε να βγουν από αυτή την κρίση. Δεύτερο ερώτημα, πολύ συγκεκριμένο. Πριν από λίγες εβδομάδες συζητήσαμε τις συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Συμβούλιο τη συζητήσατε. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα εγκάρσιο θέμα, οριζόντιο, που επανέρχεται σε διάφορα κράτη-μέλη και αυτό είναι η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Η Κομισιόν έκανε πάλι μεγάλε δηλώσει για την αύξηση της ηλικία και συστηματικά στο Συμβούλιο γίνονται συζητήσεις με άλλο τρόπο για την πρόορη συνταξιοδότηση, για την πραγματική ηλικία, αλλά τι γίνεται με την, την νόμιμη, τη διανόμου επιβαλλόμενη ηλικία συνταξιοδότησης. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δημογραφικές αλλαγές. Να το καταλαβαίνουν τα κράτη-μέλη αυτό και να το αντιμετωπίζουν. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα και ότι το Συμβούλιο αλλάζει εκεί κάπως τις συστάσεις αναχώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τα δύο μεγάλα έργα που προχωρούν στην Ευρώπη υπό την ηγεσία του Συμβουλίου Εκοφήν είναι η Δημοσιονομική Ένωση και η Τραπεζική Ένωση. Η Τραπεζική Ένωση έχει κάποια ζητήματα και προχωρούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου ε, είχαμε την οδηγία υπαριθμών 4 για τις κεφαλαιακές απαιτήσει και τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό πρότεινε το Κοινοβούλιο. Και η μεγάλη δουλειά που απομένει τώρα να γίνει είναι το σύστημα ε, διάλυση εκαθάρισης των τραπεζών. Δεν συμφωνήσαμε Περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Γενικά υπάρχει συνένεση για τα βασικά ζητήματα, αλλά εκκρεμούν ακόμα ορισμένα που θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ε, είμαστε όμως αισιόδοξοι. Θα συζητήσουμε απόψε ε, αυτό και σε διμερείς ε, συνομιλίες την Τετάρτη ε, συνεδριάζει το Συμβούλιο και θα παραμείνουμε όσο καιρό χρειαστεί, ακόμα και μέχρι αργά για να συμφωνήσουμε. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουν ε, καλή πρόθεση να βρεθεί μια συμφωνία. Για το θέμα της μεταρρύθμισης των συντάξεων, ε, σε διάφορες χώρες έχουν μεταρρυθμιστεί τα συστήματα, ενώ άλλες χώρες που είναι σε προγράμματα έχουν πάρα πολύ ισχυρή εντολή. 68 ε, θα είναι στη χώρα μας ε, και ε, οι περισσότερες χώρες έχουν τέτοια τις προτάσεις και ακολουθούν. Δεν υπάρχει δηλαδή πανευρωπαϊκά κάποια νόμιμη ηλικία οπωσδήποτε ίδια για τη συνταξιοδότηση. Και αυτό έχει νόημα κατά την άποψή μου γιατί η δημογραφία δεν είναι παντού η ίδια. Και μπορεί να είναι βιώσιμη η ηλικία συνταξιοδότηση σε μια χώρα ενώ σε μια άλλη να μην είναι. Πάντα χρειάζεται μια ισορροπία ε, ανάμεσα στο ποιο είναι το σωστό μέτρο για ε, το κέντρο ή, για ε, ε, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και η αύξηση του ορίου ηλικίας είναι κάτι το οποίο ε, τελικά θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών ανάλογα με τη δημογραφική τους πραγματικότητα. Τώρα η πράσινη, ο Φίλιππος Λάμπερτς. Καλώς ορίσατε κύριε Νούναν. Πρώτον, η Ιρλανδική Προεδρία ήταν πράγματι προεδρία που επέτυχε μερικά πράγματα Θυμάμαι το CRD4 που το επεξεργαστήκαμε και μαζί ή τουλάχιστον καταλήξαμε μαζί. Φυσικά μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τις τράπεζες αλλά τουλάχιστον υπήρξε κάποια πρόοδο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό. Ήταν πολύ επαγγελματική προεδρία και ελπίζω και άλλοι να σας μιμηθούν. Τώρα, το πρόβλημά μου είναι το BRD που λέμε. feeling as to uh, uh, what the key issues that are on the table and uh, the, the possibility of. Η τράπεζα Bert ανασυγκρότηση. Πρέπει να πω ότι με εκνευρίζει λίγο το ότι μερικοί αναφέρουν την Ιρλανδία όσα μία από τις φτωχότερε και πιο προβληματικές χώρες της Ευρώπης, αλλά άμα δω τους αριθμούς διαπιστώνω ότι μέσα στη χώρα εκείνη ο πληθυσμός έχει αντιμετωπίσει πολύ σκληρή μεταχείριση καθόλου δίκαια κοινωνικά. Στην Ιρλανδία δεν είμαι σίγουρος ότι οι πλουσιότεροι φέρουν τα μεγαλύτερα βάρη της ανάκαμψης και δεύτερον θα έλεγα ότι η Ιρλανδία πληρώνει παραπάνω από ό,τι έπρεπε γιατί δεν έγιναν μόνο δανεισμοί στην Ιρλανδία ανεύθυνοι αλλά και δανειοδοτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια για την Ιρλανδική Προεδρία ιδιαίτερα δε για την πρόεδρο στο θέμα του CRD 4. θα γνωρίζετε ότι δεν τα πετύχαμε όλα την περασμένη Παρασκευή στο Λουξεμβούργο. Παραμένουν ακόμη εκκρεμή μερικά προβλήματα και με το χρόνο που είχαμε δεν μπορούσαμε να τα λύσουμε όλα. Το θέμα ήταν μάλλον η έλλειψη χρόνου παρά οι αντιθέσεις θέσεων. Γι' αυτό λύσαμε τη συνεδρίαση και είπαμε ότι θα τα ξανασυζητήσουμε. Ελπίζω να τα βρούμε. Ως Προεδρία κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βρεθεί μια λύση και σχεδόν πετύχαμε συμφωνία. Το κυριότερο θέμα ήταν η εξισορρόπηση μεταξύ εκείνων που ήθελαν περισσότερη ευελιξία και των άλλων που ήθελαν περισσότερη εναρμόνιση. Αλλά η βασική αρχή ήταν bail-in μάλλον παρά bail-out. Αλλά μερικές χώρες ήθελαν οπωσδήποτε τη χρήση της περίπτωσης bail-out αντί bail-in. Η κυριότερη ομάδα κινήθηκε προς τον bail Ανώ μερικές χώρες, εκτός του ευρώ κυρίως, ήθελαν μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση μέτρων bailout με χρησιμοποίηση έλεγαν δικών τους ταμείων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε η συζήτηση και επεξεργαζόμαστε τώρα συμβιβασμούς. Πρέπει να δοθεί κάποια ευελιξία και η συζήτηση αφορά βασικά το βαθμό ευελιξίας που θα εγκριθεί τελικά. Αυτά θα τα δούμε την Τετάρτη ελπίζω να συμφωνήσουμε τότε. Ότι η Ιρλανδία είναι λέει το θετό παιδί των προγραμμάτων διάσωσης. Κοιτάξτε αυτό χειροτερεύει, εκνευρίζει τους Ιρλανδούς και τους λυπεί, ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για τον κόσμο και δεν είναι αλήθεια ότι δεν θυσιάζουν μερικοί. Όλοι κάνουν θυσίες στην Ιρλανδία και αυτοί που κάνουν τις περισσότερες θυσίες είναι όσοι έχασαν τη δουλειά τους. Αυτοί που έχουν δουλειά φορολογούνται κατά 52%. για ένα ζευγάρι 38.000 το χρόνο δηλαδή. Άμα τα μεταφράσετε αυτά σε ολόκληρη την κλίμακα καταλαβαίνετε ότι για όλους είναι δύσκολα. Ναι μεν είναι διαφορετικές οι προοπτικές του καθενός αλλά όλοι ζουν δύσκολα. Πάντως θα καταλήξουμε, θα πετύχουμε το στόχο του 3% μέχρι το 15%. Εδώ μιλάω τώρα ως Υπουργός Οικονομικών και όχι ως Προεδρεύων. Σημειώσαμε ήδη ένα χρόνο συνεχούς ανάπτυξης και ελπίζω να συνεχίσει αυτό. Αλλά δεν ήταν εύκολα για κανέναν και θέλουμε τα βάρη να κατανεμηθούν ισότιμα. Διατηρήσαμε τις βασικές εισφορές χωρίς περικοπές στα κοινωνικά. Όσοι έχασαν τη δουλειά τους λοιπόν είχαν τουλάχιστον κάποια επιδόματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Τέρχο από την ΕΦΤ. E Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να θίξω κάποια πράγματα που, που ήδη αναφέρθηκαν εδώ. τελευταίο, στο τελευταίο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ δόθηκαν οδηγίες για κάποια κράτη όσον αφορά την, τα ελλείμματα και τα μνημόνια. Εσείς τι πιστεύετε, πιστεύετε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί πιστεύετε, και ποιο είδους αιτιολόγηση βλέπετε για αυτήν την ε, αναθεώρηση. Κοιτάξτε, εμεί αναλάβαμε την κυβέρνηση στην Ιρλανδία το 2011 και η Τρόικα που ήταν στην Ιρλανδία τότε και είχε υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν υπό εξέλιξη. Εμεί ε, κάναμε διάφορε κυλιόμενε διαπραγματεύσει για αυτό το πρόγραμμα και η πρώτη αναδιαπραγμάτευση μα έδωσε ένα παραπάνω χρόνο μεταξύ άλλων για να φτάσουμε τους στόχους του ελλείμματος. Το πρόγραμμα ήταν ε, μέχρι το 2014, τώρα το έχουμε και μέχρι το 2015. Η δικασία υπερβολικού ελλείμματος σε διάφορες χώρες δόθηκε παραπάνω χρόνος για να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές. Τώρα που ήμασταν εμείς οι πρώτοι που πήραν παραπάνω χρόνο, ε, δεν μπορούμε να δίνουμε και μαθήματα στους υπόλοιπους επειδή ε, τους χρειάζεται παραπάνω χρόνος για να διορθώσουν την κατάσταση. Τώρα από μακροοικονομικής άποψης ε, με το Ιρλανδικό μου ιδιότητα ε, είναι το εξή. Το δικό μας πρότυπο για θέσεις και για ανάπτυξη και για να επανέλθουμε στο mainstream της οικονομικής πρόοδου το το μοντέλο μας είναι η ανάπτυξη με βάση τις εξαγωγές. Άμα οι πελάτες μας δεν αγοράζουν από εμάς δεν μπορούμε να εξάγουμε. Και αν η ζήτηση περιορίζεται σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και δεν μπορούν να αγοράσουν όσα παραδοσιακά αγόραζαν, ε, έχουμε πρόβλημα. Από τη δική μας προοπτική λοιπόν, από την Ιρλανδική προοπτική, αν κάποιες βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν παραπάνω χρόνο να προσαρμοστούν διότι και διατηρούν τη ζήτηση αλλά χωρίς να δημιουργείται παραπάνω σοκ, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν παραπάνω διορθώσεις. Είναι λεπτό το θέμα για το πώς κανείς θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να φτάσει σε έλλειμμα κάτω από το 3%. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη το 2002 είχαν ε, ήδη παραβιαστεί οι κανόνες οι οποίοι δεν ε, πανεπευλήθησαν. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι κοινοί δημοσιονομικοί κανόνες θα εφαρμοστούν και αυτό που αναζητούμε δεν είναι αλλαγή κανόνων αλλά αλλαγή του χρονοδιογράμματος εντός του οποίου ε, επιτυχάνονται οι στόχοι. Κύριος Μάρτιν. <coughs> Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση στραμμένη προς το μέλλον μάλλον. Αυτό το Σαββατοκυριακό και ε, η Αμερικανική ΦΕΔ και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών δώσανε μηνύματα σαφέστατα ότι έχουν μάλλον παρέλθει οι καιροί του φτηνού χρήματος που κατέκλυζε τις ε, αγορές και φάνηκε ε, ότι πολλές χώρες δεν κατάλαβαν, δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που τους δόθηκε με την επιμήκυνση ούτε για το χρέος, ούτε για την εξυγίαση των τραπεζών τους, όσο θα επιθυμούσαν ορισμένοι. Δεν μιλώ για την Ιρλανδία εδώ, αλλά θα με ενδιέφερε γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, είπατε ότι έχετε εδώ για τρίτη φορά, είναι η τρίτη σας προεδρία ε, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείξετε ένα νυφάλιο βλέμμα στο μέλλον για να μας πείτε πώς ερμηνεύετε αυτές τις δηλώσεις που δεν είναι τυχαίες και ταυτόχρονα είδαν το φως της δημοσιότητας. Τι σημαίνει αυτό για το επόμενο διάστημα. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όταν είχα έρθει τον Γενάρη και σας μίλησα, το παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο ήταν σε δύο φάσεις. Κίνα και ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες αφενός με ταχύς ε, ρυθμούς ανάπτυξης γενικά και τον υπόλοιπο κόσμο, τις παλιές ανεπτυγμένες οικονομίες τις είχατε σε ύφεση. Μετά από έξι μήνες έχει αναστραφεί το μοντέλο. Βλέπουμε τις αναδυόμενες οικονομίες και την Κίνα να προχωρούν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, βγήκαν από την ύφεση και τώρα αυξάνονται με ποσοστό 2,5% και 3% ετησίως. Ε, συμπέρασμα τα μέτρα που εισήγαγε η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, τα έκτακτα μέτρα, ε, και βασικά κόβουν χρήμα, όπως και να το βαφτίζουν, έχουν ε, σταματήσει σιγά σιγά να ισχύουν. Ενώ ο υπόλοιπο κόσμος και η Ευρώπη παραμένει σε ύφεση. Ε, νομίζω ότι οι Αμερικανοί φίλοι μας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους επηρεάσουμε, να, θα πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω προς την κανονικότητα στα νομισματικά, όχι με απότομες σπασμωδικές κινήσεις, γιατί αυτό θα μας προκαλέσει μας πολλά προβλήματα. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Βέβαια, ξέρω ότι δεν έχει ε, ενταλή να κάνει τα ίδια με εκείνα που κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας ή η Αμερικανική Fed ε, ε, στην νομισματική πολιτική. Ο κύριος Ντράγκη είναι και ικανός αλλά και λεπτός στους χειρισμούς του και μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει. Ξέρει ότι οτιδήποτε πράγματι θα έχει μεγάλες συνέπειες. Και το θέμα του OMT, ε, των οριστικών νομισματικών συναλλαγών, ε, θα πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά από ό,τι οι Αμερικανοί. Πάντω, καλωσορίζω το γεγονό ότι σιγά σιγά βγαίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε από την ύφεση, αλλά θα παρακαλούσα του φίλου μα, του Αμερικανού, να μην κάνουν στην πολιτική του ε, ξαφνικά άλματα, αλλά να προχωρούν με αργού ρυθμού και ομαλού. Κοιτάξτε τι γίνεται και στην Ιαπωνία. Γιατί γίνεται και μια απόπειρα να φέρνουν ένα νέο μοντέλο που δεν το έχουμε δει στη δική μας γενιά και ελπίζω αυτό να μην οδηγήσει σε αντίπεινα και μέτρα ε, ε τίμησης ε, του νομίσματος για λόγους ε, ανταγωνιστικούς. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε γενικότερα στο G7 ή στο G8 και όχι αμυγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κινούμεθα σε ένα ευρύτερο χώρο. Πάντω, εμεί θα πρέπει να εξακολουθήσουμε στο δρόμο μα στι Ευρώπη, έλεγχο του χρέους, έλεγχο του ε, λίματος, αλλά και μια στρατηγική για θέσεις εργασίας και ε, μεγέθηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Στην Ευρώπη συνήθω ισχύει ένα δημοκρατικό κέντρο. Η Ευρώπη κυβερνάται στο κέντρο. Καμιά φορά κέντρο δεξιά, καμιά φορά κέντρο αριστερά. Ε, η ανεργία των νέων σε ορισμένε χώρε έχει φτάσει στο 40 και 50% και δεν νομίζω ότι θα επιτρέψει στο μοντέλο αυτό να επιβιώσει. Και για λόγου ευρύτερου πέραν των οικονομικών νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επανακινήσουμε τις οικονομίες μας στην Ευρώπη, ε, ιδιαίτερα προς όφελος των νέων. Ευχαριστώ. Ο Βέρνερ Λάγκεν Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Στο εξάμεινο της Προεδρίας σας, όντως, είχατε πολλά δύσκολα ζητήματα να αντιμετωπίσετε στην ημερήσια διάταξη και υποχρεωθήκατε επίσης να καλύψετε και ε, αυτά που κληρονομήσατε από την Κυπριακή Προεδρία. Αναγνώριση σας αξίζει και την έχετε, αλλά παραμένουν εκρεμή ζητήματα. Μόλις μιλήσατε για την Ιαπωνία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ότι η υψηλή χρέωση και ε, η μη εξυγίανση του τραπεζικού τομέα το 1997 δεν επέτρεψαν θετικές εξελίξεις επί μία 15 ετία και ορισμένοι πρεσβεύουν αυτά τώρα για την Ευρώπη. Κάτι που δεν λειτουργήσε στην Ιαπωνία και ουσιαστικά πέτυχε επί 15 χρόνια. Θέλουν ορισμένοι να το μεταφέρουν εδώ. Να ε, αναφερθώ σε δύο σημεία που μιλήσετε κι εσείς γι' αυτά. Καταφέραμε να προχωρήσουμε, να βάλουμε μια οροφή ανάμεσα ε, στη τράπεζα και στα χρέη των κρατών. Δεν νομίζω. Η Κεντρική Τράπεζα ε, δανείζει φτηνά και ε, δεν επωφελούνται οι επενδύσεις, η ιδιωτική οικονομία, οι πελάτες, αλλά αυξάνεται το κρατικό χρέος. Αγόραζαν κρατικά ομόλογα και αυξάνεται έτσι και η εξάρτηση, δεν μειώνεται καθόλου. Και ένα δεύτερο είναι Ε, μιλήσατε για 16 νομοθετήματα, νομοσχέδια που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας ε, ε, αντιμετωπίστηκαν και πολλοί ολοκληρώθηκαν. Ακούμε όμως κατηγορίες και αιτιάσεις από τον τραπεζικό τομέα ότι είναι υπερβολική ρύθμιση ασίδωτη. Έχουμε ακούσει μάλιστα και για τσουνάμι ρυθμίσεων. Έχουν δίκιο νομίζετε και οι τράπεζες. Η εξάρτηση των κρατών από τις τράπεζες Φαίνεται και από αυτό ότι ιδιαίτερα σε μικρά κράτη, και δεν αποτελεί εξαίρεση εδώ Ιρλανδία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Μάλτα κλπ. Σε σχέση με το ΑΕΠ, ο τραπεζικός τομέας είναι και ήταν υπερβολικός, υπερμεγέθης και ξεχυλωμένος. Και μας είπατε ότι στις Ηνωμένε το 90% χρηματοδοτείται ε, στις επενδύσεις εκτός τραπεζικού τομέα. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μπαρνιέ είπε ότι θέλει να κάνει μια έκθεση για τις παρατράπεζες. Και ακριβώς αυτός ο τομέας που δεν ελέγχεται είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Πώς βλέπετε αυτή τη σύνδεση και αυτή τη σύγκριση. Όσο και σας αξίζουν έπαινοι, γιατί πολύ καλά φύγει η Προεδρία σας. Για το θέμα της Ιαπωνίας, πέρασαν 20 χρόνια με αποπληθωριστική οικονομία. Μειούμενη ανάπτυξη και παρακμάζοντα πληθυσμό. Οπότε οποιαδήποτε κυβέρνηση με εντολή να κάνει αλλαγές έπρεπε να κάνει τρομερές αλλαγές και ελπίζω τα όσα κάνουν να δουλέψουν. Αλλά τα επίπεδα χρέους στην Ιαπωνία δεν συγκρίνονται με τις Ευρώπης. Τελευταία φορά που το κοίταξα Νομίζω ότι ήταν 225% ε, του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 93-94%. Δεν είμαστε σε φάση όπου θα φτάσουμε σε αστρονομικά επίπεδα όπως στην Ιαπωνία. Και ελπίζω ότι αυτά που προσπαθεί τώρα η Ιαπωνία θα λειτουργήσει, γιατί ό,τι δοκιμάστηκε παλιότερα, λειτουργήσε και για τον ε, ορισμό τώρα των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν προκαλέσει πολύ δυστυχία στους απλούς ανθρώπους ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη και νομίζω ότι μας απογοήτευσαν ε, οι τραπεζίτες μας. Αλλά υπάρχει, έγινε μια κίνηση στις, στα τέλη της δεκαετίας των 90 στην Ευρώπη ολόκληρη και μας χτύπησε και στην Ιρλανδία και ήταν το light touch regulation, δηλαδή το να θεσπιστούν κάποιες αρχές που θα ακολουθούσαν οι τραπεζίτες, ε, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εκείνος ο κανονισμός light touch, δηλαδή ρυθμίσεις light ήταν αποτυχία. Και γι' αυτό είναι καλό που τώρα η Ευρώπη στρέφεται σε πιο αυστηρούς κανονισμούς για τις τράπεζες και νομοθεσίες. Το στηρίζω απόλυτα και πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πιστεύω πως εμείς στην Ευρώπη δίνουμε μεγάλη έμφαση στο τραπεζικό σύστημα και ότι αυτό είναι ο μόνος πόρος ε, ρευστότητας και επενδύσεων και γι' αυτό και Κατά τη διάρκεια ε, ε, της Προεδρίας μας φέραμε, συγκεντρώσαμε επιστήμονες για να διερευνήσουν τις δυνατότητες μη τραπεζικών επενδύσεων. Ως τμήμα του σχεδιασμού μας, για παράδειγμα, για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Υπουργείο μου, τον περασμένο Δεκέμβριο, έκανε ένα σεμινάριο όσον αφορά ε, τις μη τραπεζικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης και έχουμε καταθέσει τα απορίσματα στην Κομισιόν και αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομάδας. για να προωθήσει τις μη το μη τραπεζικό δανεισμό και την ε, κινητοποίηση της βιομηχανίας και των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φυσικά θα πρέπει να ρυθμίζεται, αλλά θα πρέπει να δοθεί και χώρος ώστε να ωφεληθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και να δημιουργηθεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Αντολίν Σάντσες Πρεσέντο από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Υπουργέ για την άσκηση της Προεδρίας και νομίζω πως συμβάλλατε πολύ θετικά, σε, ιδιαίτερα για κάποια από τα θέματα τα οποία προχώρησαν, όπως η οδηγία για τις τα ενυπόθηκα δάνεια. Να ευχαριστήσω την ε, ε, Ιρλανδική Προεδρία που προετοίμαστηκε πολύ καλά για το θέμα και με επικοδομητικό πνεύμα. Όμως υπάρχει ένα θέμα που παραμένει εκρεμές και που με ανησυχεί. Γιατί στον τρίλογο, το τριμερή διάλογο του Απριλίου μιλήσαμε για το άρθρο 28, το οποίο αφορά το διαθεσμικό χαρακτήρα, το διοργανικό χαρακτήρα και θα ήταν καλό να επιληθεί με οριζόντιο τρόπο. Έτσι, επίσης συμφωνήσαμε για μια άλλη οδηγία για την αρχή των πινάκων συσχέτυχης, η αντιστοιχίας για την ε, οδηγία για τις κεφαλαικές απαιτήσεις 4 συμφωνήσαμε για μια, οδηγία, μια διαδικασία να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την ενημέρωση όταν χρειάζεται πολύ εκτενής προφόρηση και επίσης είπαμε ότι χρειάζεται να σκεφτούμε κάποιο μέτρο γιατί είναι περίπλοκο το θέμα. Οι διάφορες μορφές των υποθηκών διαφέρουν αναχώρα. Επίσης αναφορά στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που είναι επίσης ε, τους κανόνες, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Στις 20 Μαΐου κρίθηκε ένα κείμενο στη μόνιμη αντιπροσωπεία. Δεν είχε όμως την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε αυτά που ζητούσαμε εμείς. Και μια οδηγία που ε, συζητήθηκε σε τριμερή διάλογο και σε τέτοιο βάθος, Πώς είναι δυνατόν να πάει σε δεύτερη ανάγνωση αν δεν ληφθούν μέτρα και θα καθυστερήσει προφανώς την έγκριση σε μια αγορά που είναι τόσο ευαίσθητη και μπορεί τόσο πολύ να βοηθήσει αν περάσει. Και μάλιστα και την ανάπτυξη σε ορισμένα κράτη της Ένωσης. Θα σας παρακαλούσα γιατί δεν τέλειωσε ακόμα η Προεδρία σας και επειδή θα συνεχίσετε να είστε συνδεδεμένοι και με το τρίο με την επόμενη Προεδρία θα σας παρακαλούσα να μην το μπλοκάρετε αυτό το θέμα και να εργαστείτε με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα για να ε, ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. Και αν μπορούσατε ε, να μας σχολιάσετε λίγο για το πώς θα αντιμετωπίσετε τα θέματα της άμεσης κεφαλαιοποίησης με αναδρομική ισχύ. Um, just before the minister replies... Αν και χρησιμοποιήσατε ε, την έκφραση πίνακες συσχέτισης, σημαίνει ε, για προσθήκη επιπλέον πληροφοριών όταν κάτι δεν είναι σαφές. Αυτό ζητά. Ε, είναι ένα άρθρο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκει αντίσταση από το Συμβούλιο, αλλά είμαι βέβαιος, γνωρίζω την, είμαι βεβαίω ότι γνωρίζω την απάντηση που θα ακούσουμε. Ναι, προσωρινή συμφωνία επί του θέματος αυτού επιτεύχθη στο τελευταίο τριμερή διάλογο στις 22 Απριλίου και η προτινόμενη οδηγία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο μέσω των πρέσβεων των κρατών μελών σε συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων στις 8 Μαΐου. Και ως εισηγητής θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω πάρα πολύ για την μεγάλη πολύτιμη σας βοήθεια το επόμενο φάση σε αυτή τη δικασία είναι το Κοινοβούλιο να ψηφίσει στην Ολομέλεια για το συμβιβαστικό κείμενο που έστειλε η Κορεπέρ με τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή Έκονα. Αυτή η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο υπό τη Λιθουανική Προεδρία. Τώρα, Επιστήνω την προσοχή σας σε ένα, επιστήσατε μάλλον την προσοχή μας στο επεξηγηματικά έγγραφα ε, και ένα σημείο όπου το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στη διοργανική συμφωνία ώστε να εξασφαλιστεί μια ομαλή πρώτη ανάγνωση και συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτής, αλλά είμαι βεβαίω ότι η επερχόμενη η Λιθωνική Προεδρία που θα γνωρίζει τις σημερινές μας συζητήσεις και το θέμα που αναφέρατε είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το γνωρίζουν. Σας ευχαριστώ. Τώρα εξ ονόματος του ΕΛΚ ο κύριος Φέιο. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επαγγελματικότητα με την οποία ασκήσατε την Προεδρία του Συμβουλίου. όπως άλλωστε και άλλες ε, προεδρίες που προηγήθηκαν. Τώρα, κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου υπήρξε μια, μια διαμάχη που αφορούσε ακριβώς ε, τα ε, προγράμματα προσαρμογής. Εγώ προέρχομαι από την Πορτογαλία και η χώρα μου προσπαθεί για να βγει από αυτό το πρόγραμμα βοήθειας ε, και προσαρμογής μέσα στο προβλεπόμενα χρονικά ωρία και θα ήθελα να γνωρίζω η Ιρλανδία πέρα, να μας πει την εμπειρία της με ποια ανάλυση κάνει για τα προβλήματα προσαρμογής τα οποία έχουν καθοριστεί. Σε τι μπορούμε να τα βελτιώσουμε, ποιες επικρίσεις μπορείτε να μας κάνετε. Ας πούμε στην ε, Πορτογαλία εμείς έχουμε τηρήσει τα κριτήρια του προγράμματος. Υπάρχουν ε, έκτακτα θετικά στοιχεία γιατί έχει μειωθεί το διαρθωτικό έλλειμμα το δημόσιας οικονομίας μας, έχει, έχουν βελτιθεί οι εξαγωγές μας, όμως ταυτόχρονα υπάρχουν επιπτώσεις στην ύφεση που αυξάνεται κάθε χρόνο και στην ανεργία που έχει φτάσει από το 12% στο 25% και όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται μια αβάσταχτη κοινωνική κατάσταση. Εσείς ποια ανάλυση κάνετε από αυτών των προγραμμάτων και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Επίσης υπήρχαν ε, Συγκρούσει ή όχι σε σχέση με τη συμμετοχή του Διεθνού Δομισματικού Ταμείου σε αυτά τα προγράμματα. Ε, ε, Εσεί θεωρείτε ότι ήταν θετική η συμμετοχή του στα προγράμματα προσαρμογής ή μήπω θα έπρεπε να ισχύσει κάποιο μοντέλο που το Δούνο του δεν θα είχε καμία ανάμειξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Και πάλι ως Ιρλανδός να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με την Πορτογαλία. Έχουμε πολλές κοινέ εμπειρίε και το είδος των όρων που συνοδεύουν τα προγράμματα ήταν κοινά. Ε, ήταν κοινή μάλλον ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Εσείς ε, υποφέρετε από τις ίδιες του ίδιου όρου όπω και εμεί, αλλά πιστεύω πω ήταν απαραίτητη. Ε, προσαρμογή του προγράμματος. Πιστεύω πως οι ε, ανακοινώσει για την, το πρόγραμμα από την πλευρά της Τρόικα θα ήταν καλές. Δημιουργήθηκαν ε, αγωνίες και προβληματισμοί μέσω της ανακοίνωσης των προγραμμάτων στα αρχικά στάδια και μόνο όταν ε, δημιουργήθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Τρόικα καθώς και τους ε, υπουργούς ε, ή τους ανώτατους υπαλλήλους μπόρεσε να υπάρξει μια πιο εύκολη ροή στην επικοινωνία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν σημαντικό σε αυτά τα προγράμματα γιατί έχουν παγκοσμίω τεράστια εμπειρία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τέτοια εμπειρία όσον αφορά προγράμματα διάσωσης και λειτουργούν και ως αντίβαρο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά του τομεί όπου η ΕΚΤ έχει εμπειρία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνει το δυνατό στα προγράμματα, αλλά ελπίζω ότι οι χώρες υπό μνημόνια θα μπορέσουν να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά και καθώς μετακινούμεθα σε διαφορετικά μοντέλα οικονομίας όπου δεν θα περνάμε από την άνθηση στην ύφεση, από τις περιοδικές ε, φούσκες να έχουμε ε, μια δηλαδή στέρεη οικονομία που θα βασίζεται στο κόστος, στην οικονομία, την πραγματική, στις επενδύσεις, στις, ε, στην, ε, στην παιδεία, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη νέων μοντέλων, σύγχρονων βιομηχανιών και κλάδων που θα οδηγήσουν ε, τον κόσμο στην επόμενη γενεά και θα ήθελα όλα και περισσότερο η Ευρώπη μέσω των πολιτικών της να αποφεύγει τα μνημόνια στο μέλλον και όχι να προσπαθεί <laughs> να σχεδιάσει καλύτερα μνημόνια. Ευχαριστώ πολύ. Γκούναρ Χόκμαρκ. Αν δεν το γνωρίζετε, είναι και ο συγητής μας για την οδηγία BRRD την ανάκτηση και την εκαθάριση τραπεζών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την περιγραφή των επιδευμάτων της Προεδρίας σας. Δυστυχώς βέβαια δεν κατορθώθηκε να επιτευχθεί πλήρης απόφαση την περασμένη Παρασκευή. Ελπίζουμε αυτή την εβδομάδα να αποφασιστούν και τα υπόλοιπα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε υπάρχουν να βρεθεί μια λύση για το θέμα όπως λέτε της ευελιξίας. Δεν θα ήταν σωστό νομίζω να πούμε ότι υπάρχει διαφορά από αυτού μεταξύ χωρών Ευρωζώνης και εκτός. Γιατί το θέμα είναι πώς θα διασφαλίσει κανείς ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που υπάρχουν σε μια χώρα μέλος πριν αρχίσει το πράγμα να γίνεται πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Επίσης δεν είναι αντίφαση μεταξύ bail-in και bail-out, διότι το εργαλείο του Μπέιλιν είναι πολύ σημαντικό και θα, στο μέλλον θα αποδειχθεί ακόμη σημαντικότερο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, καταστάσεις όπου δεν βοηθάει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί μπορεί έτσι να καταστραφεί η οικονομία ακόμη περισσότερο. Είναι λοιπόν το θέμα να έχουμε όλες τις ευκαιρίες και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας ώστε η κάθε κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ότι θα σταθεροποιήσει την οικονομία της. Στο Κοινοβούλιο καταφέραμε αυτή την εξισορρόπηση νομίζω. Δεν λέμε ή το ένα ή το άλλο. Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε και όταν δεν αρκεί να γίνονται αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις που έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι ο δρόμος για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Όχι πάντα θετικά βέβαια γιατί πρέπει να υπάρξουν και κριτήρια για τον τρόπο εφαρμογής αυτών των δημοσίων παρεμβάσεων έτσι ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων να διασφαλιστούν. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου πριν από την Τετάρτη και το ερώτημά μου είναι θα το κάνετε. Δεν διαφωνώ με την ανάλυση σας και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τα επιχειρήματά σας. Ο ρόλος της Προεδρίας σε τέτοια θέματα είναι να είναι ο ένας έντιμος διαμεσολαβητής και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ταυτίσει τον χώρο που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών ώστε η επιλογή του bailout να επιτραπεί καθώς και του bail-in στις ανάλογες περιπτώσεις. Εκεί πρέπει να, βρεθεί, να επιτευχθεί ο συμβιβασμό. Αλλά αν βασιστούμε στις αρχές, όλοι γνωρίζουμε τη φράση too big to fail. Γιατί υπήρξαν τράπεζες δήθεν too big to fail, διότι ο κίνδυνος ήταν να καταστρέψουν όλη την οικονομία. Αυτές είναι οι τράπεζες που είναι too big to fail. Πώς θα περάσουμε λοιπόν από μια θέση όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα είναι too big to fail μέσω του διαχωρισμού της ε, βασικής δουλειάς των τραπεζιτών με την κερδοσκοπική ή επιχειρηματική τους. Έτσι είχαμε πει ότι θα λύσουμε τον φαύλο αυτό κύκλο, θα βγούμε από αυτόν. Και τώρα αυτό ε, αρχίζει να εφαρμόζεται. Όταν θα φτάσουμε στην πράξη σε αυτό το αποτέλεσμα. Αν μια τράπεζα πρέπει να βοηθηθεί ή να σωθεί, αντί να έρθει το υπηκό με τα χρήματα των φορολογουμένων για να τη σώσει, η τράπεζα θα πρέπει να αναδιοργανωθεί με τους δικούς της πορους Μπέιλιν λοιπόν, αρχίζοντας από τους μετόχους. Μετά όσους έχουν ομόλογα κλπ. Ξέρετε ποια είναι η ιεραρχία που έχει αποφασιστεί. Αλλά όπως λέτε κι εσείς θα μπορούσε να έρθει μια στιγμή να υπάρξει μια κατάσταση όπου η θεωρία αυτή μπορεί να καταστρέψει μια οικονομία και να μην είναι η καλύτερη λύση. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα χωρών που έχουν αυξήσει τους φόρους και έχουν τώρα πόρους που τους μάζεψαν με τον ρητό σκοπό να λύσουν το πρόβλημα των προβληματικών τραπεζών. Δεν είναι λοιπόν θέμα in και out, αλλά το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται σε χώρες που δεν είναι ιδίω μέλη της Ένωσης. λοιπόν θα προσπαθήσω για να σας απαντήσω να πετύχω ένα συμβιβασμό όπου μία εντολή Μπέιλιν όταν εξαντλείται να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ήδη οι πόροι πέρα από αυτό το Μπέιλιν. Νομίζω ότι βασικά θα υπάρξει συμφωνία από αυτού, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος. Πώς, πότε και τα λοιπά θα αργήσουμε πολύ την Τετάρτη, αλλά ελπίζω να καταλήξουμε στη συμφωνία. Agreement Ελπίζω κοντά και με εμάς. Μικροφόνο. Ε, θα σου ξαναδώσω το λόγο και δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να βρεθεί κοινή συμφωνία στο Συμβούλιο αλλά όχι μόνο κοινή, αλλά να μπορέσει να βρεθεί και μια συμβαστική λύση με το Κοινοβούλιο, όχι μόνο να συμφωνήσει το Συμβούλιο. Ε, και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τι διαφορετικέ θέσει που έχει ο καθένα και ότι η λύση και μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κατέρωθεν τους δύο συνομοθέτε. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, ε, να κατανοήσετε και τα δικά μας επιχειρήματα. Το θέμα δεν είναι bail-in ή bail-out. Θα ήταν λάθος να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν καταστάσεις όπου ανεξαρτήτως νομίσματος κάποια μέσα που στη θεωρία είναι πάρα πολύ καλά τελικά μπορεί στην ε, πραγματικότητα να είναι περιορισμένα στην αποτελεσματικότητά τους και όχι στη συστημική κρίση που είδαμε. Και δεν θα ήταν υπεύθυνο για οποιονδήποτε από εμά να αποκλείσουμε τις δυνατότητες ε, ε, των κυβερνήσεων να σταθεροποιήσουν την οικονομία τους. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο του κοινού συμβιβασμού. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη διαφορά επί της αρχής ανάμεσα στη δική σας θέση και την ε, θέση στην οποία προσπαθώ να φτάσω, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Σίγουρα και λαμβάνω υπόψη ε, την άποψή σας γιατί δεν έχει νόημα να βρούμε, να, να, να βρούμε λύσεις στο Συμβούλιο την οποία δεν θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ Σάρον. Ε, για να συνδέσω αυτήν την συζήτηση γύρω από την ε, οδηγία για την εξυγίανση και την εκαθάριση τραπεζών με το μεγάλο θέμα της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, η πρόοδος που επετεύθη στη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου των Υπουργών ε, Οικονομικών, αλλά βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, πάρα πολλά ερωτηματικά. Το ένα αφορά ακριβώς στην ε, διασύνδεση της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης με την εφαρμογή της οδηγίας για την εξυγίανση και την εκαθάριση τραπεζών. Δεν είναι σαφές ε, πότε και υπό ποιε προϋποθέσεις θα χρησιμοποιείτε αυτό το τελευταίο εργαλείο καταφυγής, όπως χαρακτηρίστηκε στο ανακοινοθέν σας. Ε, και το δεύτερο εξίσου σημαντικό ζήτημα, κύριε Υπουργέ, που νομίζω ότι αφορά ιδιαίτερα και τη χώρα σας, την Ιρλανδία, όπως και τη χώρα μου, την Ελλάδα, όπως και την Ισπανία, όπως και την Κύπρο, όπως και την Πορτογαλία, είναι αυτή η περίφημη απόφαση για την αναδρομική εφαρμογή της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης που δεν θα γίνεται συστηματικά αλλά θα γίνεται κατά περίπτωση. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το κατά περίπτωση είναι ε, επαρκές, είναι ικανοποιητικό, δεν χρειάζεται να προσδιοριστούν κριτήρια συγκεκριμένα από πριν που να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Με ποιο γνώμονα, σε ποια βάση θα αποφασίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών εάν και πότε θα ισχύσει η αναδρομική απευθείας ανακεφαλαιοποίηση εάν δεν ε, συμφωνηθούν από τώρα αυτά τα κριτήρια και ιδιαίτερα για την Ιρλανδία που ε, φιλοδοξεί και το εύχομαι ολόψυχα να βγει στις αγορές το τέλος του 2013 ε, είναι ικανοποιητικός αυτός ο συμβιβασμός. Σας ευχαριστώ. Η διαδικασία ε, που κατέληξε στη Συμφωνία των Κατονισμών για τον ESM, για το Μηχανισμό Σταθερότητας και τη δυνατότητα ανακεφαλαίωσης τραπεζών, ε, διαρκεί εδώ και κάποιους μήνες τώρα. Ήταν μια μικρή ομάδα εργασίας και τρεις φορές συζήτησαν και στο Eurogroup αυτό το θέμα για να καθοδηγηθεί η Επιτροπή να χαράξει τις γραμμές και ε, τρεις συζητήσεις συνενώθηκα και την περασμένη Τετάρτη έγινε τελική συζήτηση για το ποιες πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα γενικά ε, είναι αναγνωρισμένο ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα της αναδρομικής ισχύς και εφαρμογής να παραμείνει ε, στις κατευθυντήριε γραμμές. Υπάρχει όμως, υπάρχει η δυνατότητα αναδρομική εφαρμογής για την ανακεφαλαιοποίηση. Κατά περίπτωση όντω θα εξετάζεται και αυτό είναι το κλειδί. Και τα βασικά χαρακτηριστικά έχουν συμφωνηθεί. Οι λεπτομέρειες και οι κατευθυντήριες γραμμές θα ακολουθήσουν. Αλλά βεβαίως, όπως και σε πολλά τέτοια πράγματα, η εφαρμογή στην πρώτη περίπτωση ε, ξεκαθαρίζει το τοπίο και δείχνει πώς θα προχωρήσουμε. Το ESM δεν έχει δώσει ακόμα χρήματα για την ε, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και δεν αναμένεται κάτι τέτοιο. Το επόμενο 12 μήνο. Από εκεί και πέρα ανοίγει αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα οριστική απάντηση περισσότερη από αυτό. Είναι κάτι το οποίο προόδευσε, αλλά κατά την άποψή μου, από την ελλαδική σκοπιά, αλλά και την σκοπιά της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, προχώρησε με ικανοποιητικό τρόπο, προς ικανοποιητική κατεύθυνση. Αλλά θα δοκιμαστεί στην πράξη και θα δείξει από εκεί και πέρα. Okay, and finally, uh, for the EPP, uh, Marianne Tyson. Marianne Tyson από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, άμεση ερώτηση σε δύο σκέλη γιατί οι ερωτήσεις της κυρίας Ποδηματά με κάλυψαν 100% από το στόμα μου το πήρατε. Ε, δηλαδή και ως εισηγήτρια για τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι περνούσα από το χέρι του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει αυτό το θέμα γιατί και αυτό ήταν προϋπόθεση για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εν πάση περιπτώσει, γενικά ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ στην Ιρλανδική Προεδρία και καταρχήν να τη συγχαρώ. Τώρα το ποτήρι μπορεί κανείς να το δει μισό γεμάτο ή μισό άδειο. Ε, για μένα είναι σίγουρα μισό γεμάτο. Έχετε κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πρόοδο. Συμφωνώ με το συντονιστή μας τον κύριο Γκοζές ότι ο κόσμος πείθεται μόνο όταν βλέπει αποτελέσματα, αλλά εμεί γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα έρχονται αργότερα μόνο και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξηγήσουμε στους ανθρώπους τι κάναμε για να έρθουν τα αποτελέσματα. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με αυτά. Ως εισηγήτρια λοιπόν για το SSM ε, πρέπει να ρωτήσω, έχει εγκρίνει το ΕΚΟΦΗΝ, έχει δει ε, ποιες χώρες που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωζώνης ε, θέλουν να συμμετέχουν στο μηχανισμό ενιαίας υποπτίας ως opt-in εθελοντικά. Επίσης έχετε καμιά ιδέα για το πότε το νωρίτερο το ΕΚΟΦΗΝ θα είναι σε θέση να ε, ε, έχει κάποια συνένεση γύρω από την πρόταση που κάνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που έχουμε διαπραγματευτεί. Δεν ξέρω μήπως έχετε να μας δώσετε περισσότερη ενημέρωση από την τελευταία συνεδρίαση. Και δεύτερη ερώτηση, σε CCTB για την κοινή ενοποιημένη βάση για το φόρο των επιχειρήσεων. Ε, ε, μας ε, απαριθμίσατε ένα κατάλογο. Ξέρω ότι η Ιρλανδία δεν ήταν πάρα πολύ ένθερμη υποστηρίκτρια, ήμουν και γι' αυτό εισηγήτρια στο Κοινοβούλιο. Δεν διαπραγματευτήκαμε γιατί ήταν απλή διαβούλευση, γνωμοδοτή εδώ το Κοινοβούλιο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει στις τελευταίες συζητήσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ε, την αποφυγή επιθετικού φορολογικού ε, σχεδιασμού. Δεν διάβασα τίποτα σχετικά με αυτή την ενιαία βάση, γιατί και αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο διαφάνειας, η καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ρωτώ λοιπόν και πάλι πώς προτίθεστε να το αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο για το CCCTB. Ευχαριστώ Πρόεδρε. very Σας ευχαριστώ πολύ. Ως εισηγητρία στον ε, νέο μηχανισμό εποπτείας ε, συμβάλλατε τα μάλα για την έγκριση του. Ε, γνωρίζουμε ότι ότι η Κομισιόν προτείνει σύντομα σχετικό ψήφισμα. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός opt-in. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν μέχρι ότου ε, εμφανιστεί η πρόταση για την φοροδιαφυγή. Νομίζω πως κανένα άλλο θέμα δεν κυριάρχησε τόσο πλήρως και τόσο απόλυτα τη διεθνή συζήτηση. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά για την εφοροδιαφυγή. και την ε, φοροαπάτη. Το φόρουμ ε, τώρα για το φόρους από των επιχειρήσεων άλλαξε ε, και συνεργαζόμαστε σενά με τον ΩΣΑ για να δούμε τις προτάσεις και συμφωνούμε όλοι όπου η λύση έγκυται στη διεθνή κίνηση, εκεί όπου δηλαδή συνεργάζονται διεθνώς οι άνθρωποι, όχι προχωρά ο καθένας μόνος του. Ελπίζαμε ότι θα είχαμε συζήτηση κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας για την ε, ε, φορολογία επί των επιχειρήσεων. Υπήρχαν όμως πολλές διαφορετικές απόψεις, οπότε θα ασχοληθεί η Λιθουανική ε, Προεδρία με το θέμα για να προχωρήσει η συζήτηση γι' αυτό. Αλλά και πάλι ο Ιρλανδός θα πω ότι εμείς πολύ θα θέλαμε να γίνει πρόοδος για αυτά τα θέματα, διότι κάθε χώρα χάνει έσοδα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Σέτζικ έφτασε, Έχασες τη σειρά σου. Θέλεις να πάρεις το λόγο, είναι δύσκολο όταν γίνονται παράλληλα συνεδριάσεις. Ε, πάντως σου δώσαμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ανταλλαγή απόψεών μας. Νομίζω πως μπορείτε να διαπιστώσετε ότι πιστεύουμε πως δουλέψατε σκληρά. Απλώς ε, θέλουμε ακόμη περισσότερα. Ε, <coughs> αλλά Υπήρξαν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις αλλά και καλές και τα αποτελέσματα ήταν ε, πολλές φορές πολύ θετικά και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει το ίδιο ρυθμός και με τους διαδόχους σας ώστε να έχουμε στο τέλος της εντολής μας ε, ολοκληρώσει το έργο μας. Έτσι ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση 8 Ιουλίου στις 3 και πάλι την, Τετα... την Τρίτη στις 9 Ιουλίου στις 9 το πρωί και στις 3. Α, όχι. Δύο και μισή αρχίζουμε τη Δευτέρα για να υπάρχει αρκετός χρόνος με τον ε, Πρόεδρο της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων, για την Προεδρία σε όλες τις ε, συνεδριάσεις που προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε σε φακέλους κοινού, ε, κοινού ενδιαφέροντος. Χωρίς την εξαιρετική σου Προεδρία δεν νομίζω ότι θα είχαμε κάνει την πρόοδο αυτή όλοι. Να ευχαριστήσω και τους διάφορους εισηγητές ε, και όλα τα μέλη της ΕΚΟΝ, διότι κατά τη γνώμη μας σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς τις σχέσεις σχέσεις μεταξύ μας και τη συνεργασία μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Thank you very much. Και εμείς ευχαριστούμε.